Good morning, colleagues, petitioners, guests, and welcome to... Καλημέρα σας, αναφέροντε συνάδελφοι. καλώ ήρθατε στην πρωινή συνεδρίαση. Καθώ κάθεστε, χαίρομαι να σα ενημερώσω για τα αποτελέσματα της χτεσινή συνεδρίασης των συντονιστών, χτες το απόγευμα. Εάν μπορείτε παρακαλώ καθίστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ησυχία ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να ακούν αυτά που λέω. Πρώτα απ' όλα η, το αίτημα των ομάδων για μελλοντικέ μερικέ διατάξει. Εγκρίθηκε με κάποιες τροποποιήσεις. Κάτι πιο σημαντικό τώρα όσον αφορά την αναφορά για το Brexit. Θα συζητηθούν στις 21 Ιουνίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και τα ευρήματα της ακρόασης για τον Brexit της 11ης Μαΐου. όσον αφορά την ακρόαση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις 22 Ιουνίου. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές για το Brexit και να χρησιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο ημέρα της ημέρας για το Brexit ώστε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες. Επίσης θα ασχοληθούμε με τις αναφορές για τον Brexit του 2007. 17. Τις πρόσπατες. Κάποιες είναι πολύ πρόσπατες. Θα ασχοληθούμε μαζί της με την επίγουσα διαδικασία ώστε να τις ε, συναθρήσουμε και να είναι όλα ξεκάθαρα για την 21η Ιουνίου. Όσον αφορά τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις, Πρέπει να σας πω πως η Επιτροπή Απασχόλησης δεν συμφωνεί για την εφαρμογή του άρθρου 54 στην περίπτωση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία, αλλά όπως ξέρετε ήμασταν ιδιαίτερα ενεργητικοί στον τομέα αυτό. Οι συντονιστές μου έδωσαν την εντολή να επαναδιαπραγματευτώ με την Επιτροπή Επασχόλησης με το στόχο να εφαρμοστεί το άρθρο 54. αφού λύσαμε την σύγκρουση αρμοδιοτήτων, η απόφαση του εισηγητή αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Οι προσβαλόμενες συστάσεις εγκρίθηκαν. Αρκετά από τα σημεία έκλεισαν, κάποια έμειναν ανοιχτά. Διερευνητικές επισκέψεις και ακροάσεις. Είχαμε πολλές διερευνητικές επισκέψεις και χαίρομαι γι' αυτό όπως και για το ότι τόσο πολλοί συνάδελφοι δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτές. Η πρώτη θα λάβει χώρα στις 22 και 23 Μαΐου στην Ισπανία. Εγκρίναμε ένα σχέδιο προγράμματος και η Γραμματεία θα συνεχίσει να εξετάζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης συναντήσεων, ένταξης συναντήσεων με τις τοπικές αρχές έστειλα στην Κονφερένθια Επισκοπάλ Σπανιόλα στην Ιερά Σύνοδο της Ισπανίας μία επιστολή ζητώντα μία συνάντηση κατά την επίσκεψή μας. Εάν απαντήσουν καταφατικά, τότε η συνάντηση αυτή θα ενταχθεί επίσης στην ημερήσια διάταξη. Η διερευνητική επίσκεψη στο Ταράντο θα λάβει χώρα από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου η σύσταση της αποστολής εγκρίθηκε. Θα συμμετάσχω στην αποστολή. Η διερευνητική επίσκεψη στη Λάρνακα προτείνεται να γίνει στις 20 έως 22 Σεπτεμβρίου. Τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μελών μας επιτρέπεται με άλλα λόγια να έχουμε έξι μέλη και τέσσερις εξοφίσιο, δηλαδή συνολικά δέκα βουλευτές θα μπορούσαν να έρθουν. Θα πρέπει να υποβάλουμε τα ονόματα πριν τις 17 Μαΐου. Τρεις διερευνητικές επισκέψεις και ακροάσεις ακόμα περισσότερες. Έχουμε πολλές ακροάσεις. Στις 21 Ιουνίου η ακρόαση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα όπως σας είπα, από το μεταθέσαμε από τις 21 στις 22 Ιουνίου για να εστιάσουμε στο Brexit στις 21. Η απόφαση για το τελικό πρόγραμμα θα ληφθεί στις 3 Μαΐου στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΕΤΗ. Όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά μειονοτήτων, θα λάβει η χώρα στις 4 Μαΐου η ακρόαση για το Brexit που θα διοργανωθεί από κοινού με τη ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει στις 11 Μαΐου. Η ακρόαση για την ανηθαγένη από κοινού με τη ΛΥΝΤΕ θα γίνει στις 29 Ιουνίου και τα μέτρα για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εκεί αποφασίσαμε για μια προφορική ερώτηση ή και ένα ψήφισμα μετά την ακρόαση για το θέμα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα εμπλέξουμε και την Επιτροπή απασχόληση καθώς είναι το πεδίο αρμοδιοτήτων της. όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, εάν τα μέλη της Επιτροπής ΠΕΤΗ θέλουν να υποβάλουν προτάσεις, τότε θα πρέπει να υποβληθούν πριν την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας, δηλαδή της 29 Απριλίου. Στα διάφορα υπήρχε μόνο ένα σημείο. Η επιστολή, η απάντηση στην επιστολή μου στον πρόεδρο Ταγιάννη όσον αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 2016. Αυτά είναι όλα. Η κυρία Εύη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ήθελα απλώς να σας επισημάνω κάτι σε σχέση με την ημερήσια διάταξη της 20ης και 21 Ιουνίου. Είχαμε επιβεβαιώσει για την αναφορά 98 του 15 της σχέσης ε, Μπελίνη. Ήδη είχαμε πει ότι αυτή η αναφορά θα μπει στην ημερήσια διάταξη. Αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τις αναφορές για το Brexit. Αλλά σας παρακαλώ την αναφορά να την κρατήσετε για εκείνη την συνεδρίαση του Ιουνίου. Γιατί ε, σκεφτείτε, είναι caregiver ε, η αναφέρουσα. Δηλαδή παρέχει δηλαδή φροντίδες κατοίκων. Οπότε η κατάστασή της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε γι' αυτό σας παρακαλώ ε, να συζητηθεί τότε αυτή η αναφορά. Κύριε Πρέντα, συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά εγώ ήθελα να σας παρακαλέσω να αρχίσουμε ψηφορίες, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε και σε άλλες επιτροπές, αν γίνεται. Έχετε, έχετε δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Τότε εγώ ήθελα πρώτα να σας μιλήσω για του τονιστέ και αυτό έγινε, ολοκληρώσαμε. Για να δούμε τώρα. Για, για το θέμα που είπε να το δούμε τα στι Πάμε τώρα στι πρώτα πρώτα γνωμοδότηση για δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων για μικρές διαφορές. Ψηφίζουμε. Amendment 6 in favor. Against. 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Favor. Against. 46. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 και 47 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα ψηφοφορίες. Και εγκρίνεται. 40. 8 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 9 και 54 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος. Μη λέτε όχι, πέστε ας επαληθεύσουμε, ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε και πέρας ψηφοφορίας. Άμα δεν το χέρι σας, δεν μπορώ να διακρίνω. Και εγκρίνεται. 55, όχι, 56 διευθύνει πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται.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 δεν 16. Δεκαέξι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, όχι εγκρίνεται, διορθώνει πρόεδρος. 17 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ένα. Συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ. Α, και την, όχι την 20, και την 20 θα κάνουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 21, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέραστη ψηφοφορίας και εγκρίνεται η 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ Την 30, α, έχετε δίκιο. Πρέπει να αλλάξω γυαλιά. Δεν γίνεται δουλειά με αυτά. Υπέρ του 30. Κατά αποχές. Έλεγχος για το 30. Με σαφή, ξεκάθαρη πλειοψηφία εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 γλωσσική, 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική. Ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. E okay, so thank you to those of you that, that came only for the vote. Ευχαριστώ όσους ήρθαν μόνο για την ψηφοφορία και συνεχίζουμε. co-chair, are you not grateful for us who are here to do the work? And only for those who came, came here only for the vote? <laughs> I'm sorry. You thank those... Συγγνώμη, ευχαριστήσατε λέει η κυρία. Το αστείο είναι ευχαριστήσατε μόνο εκείνου που ήρθαν για την ψηφοφορία κυρία Πρόεδρε. Γιατί όχι όλου. Η Πρόεδρος, ναι αλλά στην αρχή της ε, συνάντησής μας καλώς όρισε τους πάντες. Ωραία. Ας περάσουμε στην αναφορά 172. Ο κύριος Μαρσέλο την έχει υποβάλει Προσφέγον και παρευρίσκεται. Πρόκειται για ε, μια αναφορά σχετικά με τις μειώσεις του ποσοστού αναπηρίας στην αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια. Αλλά πριν συζητήσουμε την αναφορά αυτή, η Ελεονόρα, είχατε θέσει ένα θέμα που έχει σχέση με ε, την αναφορά 98 του 2015. Το σημείωσε η γραμματεία, θα δω πώς μπορούμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στην ημερήσια διάταξη ε, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε το έτοιμά σας. Ε φροντίζοντας να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και στη συζήτηση για το Brexit, πάντως θα προσπαθήσουμε. Ας προχωρήσουμε τώρα στη ε, συζήτηση της αναφοράς. Καλώς ήρθατε κύριε Μαρσέλο, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. <clears throat> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, αγαπητοί διερμηνείς, προσκεκλημένοι, όλοι όσοι βρίσκεται εδώ. Θέλω να σας ε, απευθυνθώ γιατί έχουμε πάρα πολλούς που έχουν προσυπογράψει αυτές τις αναφορές την 1062 και την 172 του 14 και του 16 αντιστοίχως πρώτα πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας σε αυτή την επιτροπή που ολοκληρώθηκε με αυτό το ψήφισμα της 7ης 7 του 2016. Επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί το πόσο απευθυνθήκατε ε, στην ε, ε, διοίκηση της περιοχής της Βαλένθια. Μιλούμε τώρα για το τι γίνεται όσον αφορά τις μειώσεις ποσοστού Ε, Πρόκειται για τα όσα σας έχει διαβιβάσει η αυτόνομη διοίκηση της περιοχής. Πρόκειται για 30 σελίδες. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν το το ότι κατά 50% το 2012 και 2013 μειώθηκε ε, το ποσοστό αναπηρίας. Μιλούμε για 50% των αναπήρων που είχαν προηγουμένως κάποιο είδους περάσει από κάποιο είδους αξιολόγηση ε, προσωρινή. Και θα πρέπει τώρα επομένω να ξανααξιολογηθούν, γιατί πέσανε μία πενταετία. Αλλά έχουμε μόνο 40 μέρες σαν προθεσμία. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να σας διαβιβάσουμε τη δική μας τεχνική ανάλυση όσον αφορά κάποια συμπεράσματα της επίσημης έκθεσης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ε, δεν έχουν αξιοπιστία. Ε, πρόκειται για κακή πρακτική και κακοπιστία όσον αφορά το πώς έγινε αυτή η αξιολόγηση. Και έφτασαν μέχρι το σημείο ε, να έχουν κάποια απαράδεκτα συμπεράσματα για οποιοδήποτε ξέρει την ε, ε, επιστήμη αυτή. Φτάσανε στο 95% όσον αφορά τη, τα συμπεράσματά τους και πες κατώ των ε, δειγμάτων. Πρόκειται επομένω τώρα για την ανάγκη να υπάρξει κάποια έρευνα ανεξάρτητη που να είναι σύντονη με την νομοθεσία που ισχύει και να δούμε κατά πόσον η διοίκηση ενήργησε με τρόπο σύνομο. Επομένως θα πρέπει και εσείς να έχετε τα δικά σας συμπεράσματα όσον αφορά το πόσο σοβαρή είναι η έκθεση της διοίκησης. Με την δική μας ανάλυση ε, προσπαθήσαμε επίσης να απευθυνθούμε στην διοίκηση της περιφέρειας και θέλουμε να υπάρξει κάποιο είδους λύση στο πρόβλημα. να υποχωρήσουν και δύο πλευρές. Ε, να σταματήσει αυτή η περίοδος του άγχου της αβεβαιότητας που ήδη έχει κρατήσει πέντε χρόνια. Και στις τέσσερις του μηνός μας κάλεσε η διοίκηση. Απλώς θέλανε να μας πούν ότι θα αναστείλουν την πρόοδο των εργασιών. Ε, και αυτό αντιφάσκει σε σχέση με όσα είπανε σε εσά. Τώρα επομένως η κατάσταση έχει μπλοκαριστεί και ε, πριν από τέσσερις μήνες επίσης καταθέσαμε τα σχετικά έγγραφα στην ε, εισαγγελία της ε, περιοχής για δεσμενή διάκριση και ούτως ώστε να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία Επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εσωτερική πολιτική ε, που προβλέπει το ότι η Επιτροπή σας θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, τα όσα προβλέπει ο ΙΕ για τους αναπήρους. Και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να τύχει καλύτερη υποδοχή η αναφορά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης επισημαίνει ότι υπάρχουν τέσσερα άρθρα των ιδρυτικών συνθήκων που αφορά ακριβώς τις δυσμενείς διακρίσεις επί τη βάση του εδαφικού κριτηρίου και αφορά επίσης την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές. Και εκεί αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει. Όμως έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή σας. Οπότε ήδη τα έχουμε πει στην ε, ε, περιφέρεια, στη διοίκηση της ε, Βαλένθια και έχουμε επίσης το ψήφισμά σας, το σημείο 162, που λέει ότι ζητείται από την Επιτροπή των Αναφορών να εποπτεύσει με προσοχή τις πολιτικές και τα σχετικά μέτρα όσον αφορά τους αναπήρους. Επομένω, ε, αυτό είναι κάτι που ήδη είχε απασχολήσει δικαστικές αρχές σε Ισπανία, σε Ευρώπη, παντού. Και επίσης έχουμε αυτά τα σημεία που, στα οποία αποδίδει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ. Ξαναγυρίζουμε όμως στην αναφορά γιατί τώρα πρόκειται για ληστεία, δηλαδή μας αποστερούν το μέλλον. Πρόκειται για θεσμικού χαρακτήρα δυσμενή διάκριση, όπως λέει το γυμνό του 15. Ε, μας αρνούνται το γεγονός του ότι είμαστε ανάπηροι. Έχουμε εδώ συγγενείς των ε, θυγέντων. Ζητούμε επομένως απόδοση δικαιοσύνης και αποζημίωση. Θα πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ένας στους εκατό αναπήρους μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Γι' αυτό και κάνουμε ομαδικές αγωγές. Θα πρέπει να έχετε την ευαισθησία να αναγνωρίσετε το τι έγινε και να ε, καταπολεμήσουμε αυτή την ε, πρακτική που φύγει τους αναπήρους. Διακόπτει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σας έδωσα 5 λεπτά, μιλήσατε με 7 λεπτά και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για τα όσα μας εξηγήσατε και τώρα πάμε στον εκπρόσωπο των αρχών της Βαλένθια, τον κύριο Άλβαρες. Καλώς ορίσατε, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ. Έχουμε λάβει τα σχετικά έγγραφα και τώρα έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας πω ε, ότι χαιρετίζω τον κύριο Μαρθέλο και όσους εκπροσωπεί. Από το 2012 3 είπαμε ότι κάνουμε μια γενική αναθεώρηση των αξιολογήσεων για την αναπηρία, ούτως ώστε να αξιολογηθούν τα ποσοστά αναπηρίας και επίσης να δούμε ε, τι πλέον εκτίματα, τι βοήθεια θα δοθεί στους ε, αναπήρους. Τι συμβαίνει τώρα. Δεν έχουμε αυτονομία ούτως ώστε ανεξαρτήτως από την υπόλοιπη χώρα να έχουμε κάποια ε, κριτήρια για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ποσοστό σοβαρής αναπηρίας. Και επευθυνθήκαμε επίσης και στον διαμεσολαβητή. Και επίσης στον αρμόδιο ε, της ε, αυτόνομης διοικητικής μας περιφέρειας. Επίσης κάναμε ε, έρευνα και τον Δεκέμβριο του 2014 καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα ότι δεν προκύπτει ότι έχουν παραβλαβεί κάποια δικαιώματα, κάποιες αρχές όπως ε, περιέχονται στο Σύνταγμα και στα ιδρυτικά κείμενα της ε, διοικητικής περιφέρειας. Επίσης, στην Βουλή της Διοικητικής Περιφέρειας το Σοσιαλιστικό Κόμμα ε, έκανε κάποιο ψήφισμα σε σχέση με τις καταγγελίες ούτω ώστε να μελετηθεί κατά πόσον εδώ υπάρχει περίπτωση αποζημίωσης. Τώρα, εμείς ε, διαχειριζόμαστε τα των αναπήρων και συνεργαζόμαστε και με τη σημερινή και με την προηγούμενη κυβέρνηση της αυτόνομης διοικητικής περιφέρειας λαμβάνουμε υπόψη και σεβόμαστε τους καταγγείλαντες για να εξεταστεί το κατά πόσον δεν έγινε σωστή αξιολόγηση της αναπηρίας και από τον Ιούλιο του 2015 ξεκινήσαμε την διαδικασία για να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυσμενής διάκρισης βάρος αυτών των αναπήρων τη σχετική περίοδο. Και κάναμε πάρα πολλές ε, συναντήσεις για να δούμε τι έχει γίνει με τις αρμόδιες αρχές και επισημαίνουμε ότι πολλοί από αυτές τις αρχές, αυτούς τους φορείς μάλλον, που τώρα έχουν προσφύγει σε εσά, μας ε, διαβίβασαν αυτό το κείμενο. Και είπαμε ότι πολλοί από αυτούς τους φορείς δεν ήρθαν στις συναντήσεις που εμείς κανονίσαμε να γίνουν και είπαμε ότι πρώτα πρώτα έχουμε ε, χίλιους που έχουμε μελετήσει και δεν καταλήξαμε πουθενά. Και όσον αφορά τους καταγγείλαντες είπαμε ότι υπάρχει ζημία λένε για αυτούς τους, των οποίων το ποστό απειρίας μειώθηκε. Και ακολουθεί τώρα η διαδικασία και τελικά λήφθηκε μια απόφαση που αναγνώρισε την ζημία και άλλαξε αξιολόγηση για μόνο τέσσερις περιπτώσεις. Για αυτή την περίοδο μεταξύ του 2012-2013 είχαμε 34.100 ε, αναθεωρήσεις της αναπηρίας και είχαμε επομένω σημαντική αύξηση. Αποτέλεσμα της αναθεώρησης είχαμε ένα 14% περίπου 4.000 των οποίων έγινε μείωση του ποσοστού και πήγανε σε κατώτερη κατηγορία. Περίπου στους 1.929% ανέβηκαν όσον αφορά το ποσοστό υπηρεσίας και κέρδισαν όσον αφορά τα επιδόματα. Οπότε είχαμε έρευνα από τις υπηρεσίες μας και με αυτή την αναθεώρηση άλλο ε, έγινε μείωση, άλλο όχι. Σας λέω εν κατακλείδη ότι η γενική μας διεύθυνση συνεχίζει τις ε, επαφές ούτω ώστε να σας δώσουμε κάθε πληροφορία που θέλετε σε σχέση με ό,τι έχετε ζητήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σούμπερτ. Ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους των αναφέροντων και τις τοπικές αρχές. Αντιδράσαμε στην αναφορά στο μέτρο που μας επιτρέπουν οι νομοθετικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλος σχεδιασμός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών παροχών ως προς τις αναπηρίες αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δράσει στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που υπόθηκε ήδη σήμερα. Αυτό που κάνουμε είναι πως ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προβούν σε μεταρρυθμίσεις για να στοχεύσουν καλύτερα και να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία και οι, τα άτομα με αναπηρίες είναι μεταξύ αυτών και να τους προστατεύσουν από τις συνέπειες της κρίσης μέσω κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας. Έχουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καταδείξαμε τις ελλείψεις που έχουν υποδείξει οι πολίτες. Έχουμε λάβει πολλές καταγγελίες μεταξύ άλλων και από την Ισπανία όπου οι πολίτες παραπονιούνται <coughs> για τις γεωγραφικές ανισότητες όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας. Το καταδείξαμε αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμεινο οι εκθέσεις αναχώρα για το 2017 είναι διοριστικές και η εκθέση για την Ισπανία περιέχει τις δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις ανισότητες που υπάρχουν ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία στην Ισπανία. Επιτρέψτε μου επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρόταση που περιλάβαμε στην έκθεση. Το μερίδιο ανθρώπων που αναγνωρίζονται ως ανάπηροι, που λαμβάνουν παροχές, διαφέρει αναπεριοχή, μεταξύ λιγότερο από 70% έως 100% και μεταξύ 20% έως 100% για τον βαθμό 1. Τι κάνουμε λοιπόν, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση. Απογράφουμε όσα γράφουν οι πολίτες στις εκθέσεις, στις επιστολές τους και αυτά που ακούμε επίσης από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, από τους εταίρους μας, από ΜΚΟ και από άλλους και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με τα μέσα που διαθέτουμε. Αλλά παρακαλώ μην, ξεχνάτε την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε παρά να εργαστούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ για την ξεκαθαρή θέση σας και επίσης για τη θετική στάση σας ως προς την ενθάρρυνση των κρατών μελών να κάνουν ό,τι δυνατόν. Ανοίγω τη συζήτηση για τους συναδέλφους και θα δώσω προτεραιότητα, προτεραιότητα σε μέλη της Επιτροπής ΠΕΤΗ και στη συνέχεια θα ανοίξω τη συζήτηση και για τα μη μέλη της Επιτροπής ΠΕΤΗ. Η κυρία Αλβιόλ πρώτα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τους αναφέροντες, αναφέροντες που ήρθαν εδώ και πάλι να μας επισκεφθούν, ούτως ώστε να μας εξηγήσουν αυτή την αδικία που τους ε, έχει πλήξει και στην ε, διοικητική περιφέρεια της ε, Βαλένθια. Πάρα πολλές φορές είμαστε ουραγίοι όσον τη χώρα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Ουσιαστικά πρόκειται για μποϊκοτάρισμα του σχετικού νόμου για τη βοήθεια των αναπήρων. Ε, ε, Καθυστερήσει, ε, πάρα πολλοί ανάπηροι που έπρεπε πολλά χρόνια για να γίνει δεκτή η αίτησή τους και στη συνέχεια για να έρθει η ώρα να εισπράξουν τα επιδόματα και κάποιοι πέθαναν περιμένοντας, περιμένοντας τις σχετικές αποφάσεις. Οπότε το, το σύστημα έχει γίνει τελείως ιδιωτικό. Οπότε έχουμε αυτό το μποϊκοτάρισμα, το σαμποτάζ το χάο και επομένως αυτό μας λένε τώρα οι αναφέροντε, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χωρίς να έχουν βελτιωθεί όσον αφορά την αναπηρία υποβιβάστηκαν για το ποσό αναπηρία και άρα μειώθηκαν και οι, ε, οι, τα, τα επιδόματα. Και όλα αυτά τα είχαμε πει από την αρχή, οπότε κάποια πράγματα βελτιώθηκαν όσον αφορά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αλλά όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας δεν έγινε κάποιο είδους ε, αναθεώρηση, δεν δόθηκε κάποιο είδους αποζημίωση. Οπότε νομίζω ότι έχουν δίκιο οι αναφέροντες και επομένως η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να αναλύσει το τι έγινε, να δώσει μια απάντηση στους αναφέροντες. Μιλούμε για δυσμενή διάκριση εις βάρος αναπήρων. Μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Επομένως κάτι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να βρεθεί η αρμοδιότητα του να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε στις αρχές της περιφέρειας. Να εξετάσουν, να αναθεωρήσουν, να κάνουν ό,τι δεν έκαναν τότε. Να αποζημιώσουν και ποτέ κανείς να μην υποστεί αυτή τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας χωρίς να έχει κάποια βελτίωση στην ε, υγεία του. Και σας ξαναλέω ότι πρόκειται εδώ για αναπήρους. Thank you, Mr. Thank you. Συγχαρητήρια κύριε Μαρσέλο. Μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ καλά. Επίσης, συγχαρητήρια και στον εκπρόσωπο της Διοικητικής Περιφέρειας. Και αυτός που μας τα εξήγησε όλα, που ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα είπε. Το θέμα είναι ότι κανένας τελικά δεν ευθύνεται για τίποτα. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Τα λέει η Κομισιόν ότι εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Η διοικητική περιφέρεια λέει ότι ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος, το κράτος έχει αρμοδιότητα. Ναι, αλλά εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει κάτι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν συζητούμε περί των εφαρμοστέων κριτηρίων. Αυτό που συζητούμε είναι η εφαρμογή των κριτηρίων. Άρα δεν μπορεί κανείς να ανοίξει τα σχήρα του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η περιφέρεια. Γιατί αυτοί πρέπει να κάνουν την εφαρμογή των κριτηρίων και να κάνουν και την αναθεώρηση. Αναγνώρισαν ότι υπήρχε ένα κάποιο χάος. Υπήρξε αναρχία. Ότι δεν έγινε σωστή αναθεώρηση σε κάποιες περιπτώσεις. Πολλές σχέες και αμφιβολίες και μου φαίνεται ότι στις ε, αναθεωρημένες υποθέσεις τελικά ε, καλύφθηκαν οι διπλάσιοι από όσους δεν ε, πέρασαν από την αναθεώρηση. Οπότε 4.000 έναντι 2, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ίσως δεν έχουν τους πόρους, ίσως δεν είχαν το χρόνο ή της περιφέρειας. Αλλά θα πρέπει να δούμε το θέμα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται για κάποιους που όχι μόνο επέστησαν αυτή την αδικία αλλά είναι για ανάπηροι. Άρα οι αδικίες βάρος των αναπήρων είναι μια πολύ σοβαρή, μεγάλη αδικία. Γι' αυτό και σας λέω να συνεχίσουμε μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σίγουρα η περιφέρεια τώρα έχει φέρει κάποιες βελτιώσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις αιτίες και τα αποτελέσματα από αυτή την αδόκιμη εφαρμογή των κριτηρίων. Και να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Βαλίνα, έχει το λόγο. Και ο κύριο Τερικάμπρα και η Μαρίνα τα εξήγησαν, να μην πω τα ίδια. Αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Πρόκειται τώρα για ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό συζητάμε. Και λυπάμαι, όπως είπε και ο Τερικάμπρας ότι δεν μπορεί να είναι όλοι Μιλάμε εδώ για δεσμενή διάκριση, για ανθρώπινα δικαιώματα. Μα αυτά κατοχυρώνονται στο Ισπανικό Σύνταγμα. Είναι αντισταγματικά αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα θα ασχοληθεί η εισαγγελία. Άρα, μα είναι δυνατόν να μην ασχολούμαστε με ανθρώπινα δικαιώματα και με τι διακρίσεις. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, τότε τι κάνουμε, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Μιλάμε για τρομερή καθυστέρηση, περιμένουμε, πεθάνουν περιμένοντας κάποιοι ανάπηροι μέχρι να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Ε, αυτό είναι αφόρητο για μια, μια κοινωνία με κράτος δικαίου τον 21ο αιώνα. Να μην ανοιχτεί αναφορά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ροδρίγκης Πυρνέιρου Φερνάντες, παρακαλώ. Muchas Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να αναγνωρίσω το έργο των αναφερόντων και των άλλων φορέων που φρόντισαν το θέμα να μείνει ζωντανό. Ευχαριστούμε και την Διοικητική Περιφέρεια για την ενημέρωση. Τώρα, προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μιλάμε εδώ για ανθρώπους και όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για πρόσωπα τα οποία λόγω της αναπηρίας τους είναι πολύ ευάλωτα. Καταλαβαίνω τις αμφιβολίες για τον τρόπο που έγινε αυτή η αξιολόγηση. Πάντως, επί κυβέρνησης Λακού Κόμματος, η διοικητική περιφέρεια δεν έδωσε καμία προτεραιότητα ή στο να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία. Οπότε αξιόλογο το έργο που έχει γίνει, αλλά θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το ότι γίνανε κάποιες ενέργειες από την περιφέρεια. Να δούμε ο καθένα τι αρμοδιότητα έχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρουμε. ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Κομισιόν λόγω της επικουρικότητας. Άρα θα έπρεπε να ασχοληθεί η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές και μας είπε ο εκπρόσωπος της περιφέρειας για κάποια θέματα τεχνικά. Ότι δηλαδή η αυτόνομη κοινότητα δεν μπορεί να ασχοληθεί αλλά το κράτος. Οπότε θα πρέπει να δούμε το τι ζημία έχουν τώρα αυτά τα πρόσωπα λόγω της μη εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει να δούμε επομένως τι κριτήρια προβλέπει το κράτος και πώς τα εφήρμοσαν. Να, τι πρέπει να κάνει η περιφέρεια. Έχουμε εδώ πέρα τις καταγγελίες, έχουμε τις ε, αιτήσει και είπανε ότι από τις σχετικές καταγγελίες των ε, χρηστών, αυτή δηλαδή που πέσαν τη του ποσοστού, ήταν 1505. Σε 73% δικαιώθηκε και επίσης ε, 16% πήγανε σε ανώτερο, ανώτερη κατηγορία και 11% σε κατώτερη κατηγορία από αυτό το 27% που άλλαξαν κατηγορία. Το θέμα είναι πώς εφαρμόσαν τα κριτήρια για την αξιολόγηση και τι έγινε με το αποτέλεσμα. Ε, νομίζω ότι έγινε κάποια βελτίωση, άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η αξιολόγηση, πώς έγινε η αναθεώρηση. Όλοι θα πρέπει να περάσουν από αναθεώρηση και όχι μόνο ένα δείγμα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα. Πολύ σημαντικό. Να μην υπάρχουν σχέσεις αμφιβολίας. Εντάξει, κάποιον άλλαξε η κατάσταση. Να δοθεί προτεραιότητα και η περιφέρεια ασχολήθηκε τελικά με τις ε, αιτήσει και προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές. Θα πρέπει επομένως να λυθούν τα προβλήματα αυτά του παρελθόντος. Και τελικά ο καθένας να του αναγνωστεί το σωστό ποσοστό αναπηρίας και να πάρει τα επιδόματα που δικαιούται. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στον κατάλογο ομιλητών. Θα ξαναδώσω το λόγο λοιπόν στον αναφέροντα τον κύριο Μαρσέλο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ λέγοντας ότι συνεχίζει να υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά την νομοθεσία για την αναπηρία αφενός Τα έχουμε ξαναπεί εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Μα δεν, όχι. Ε, δεν άλλαξαν τα τεχνικά κριτήρια. Αυτό που θέλουμε είναι να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο την Ισπανία αλλά όλες τις χώρες. Και τελικά θα αποφανθεί η εισαγγελία. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Να κρυφεί το αν έχουμε δίκιο ή όχι. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε για ρητορικέ ασκήσεις, ούτε για χαρακτικισμούς. Σίγουρα δεν πρόκειται εδώ για κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Αυτό που θέλουμε είναι να προστατεύσει η Επιτροπή σας αυτό το οποίο συζητούμε, τα δικαιώματα δηλαδή των αναπήρων. Να υπάρξει ένα πλαίσιο. Δυνάμει του, αρθρου, του 33 της ε, διακήρυξης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια σε πολλές περιπτώσεις. Άρα, να κάνετε το καθήκον σας ως Επιτροπή Αναφορών, να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, ούτως ώστε να υπάρξει το φως και να πρετανεύσει η αλήθεια. Αλλά και να υπάρξει αποζημίωση. Εμείς φροντίζουμε τους ε, αναπήρους και είμαστε και ίδιοι ανάπηροι. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Α, και ήθελα να με την Τούρινματ. Το ότι είναι θλιβερό το να πρέπει κανένας για το αυτονόητο να δώσει μάχη. Έλεγε λοιπόν Τούρινματ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ταξιδέψατε και ήρθατε μέχρι τις Βρυξέλλες για να μας περιγράψετε την εμπειρία σας και τις, τα προβλήματά σας. Θα ήθελα επίσης να ε, ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Βαλένθια για την λεπτομεριακή απάντηση που μας στείλατε και για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ήρθε η ώρα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποιο σύνοψη. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ε, όπως βλέπετε τα μέλη της Επιτροπής ε, τους απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα, αντιλαμβάνονται τη σημασία του. Τώρα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Όπως εξήγησε και η εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο η αρμοδιότητα ε, είναι των αρχών της Βαλένθια. Αυτό το γνωρίζει και ο αναφέρον. Το μόνο που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εκφράσει τη λύπη του, την ανησυχία του και να ενθαρρύνει, να παροτρύνει τις Ισπανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, να αντιμετωπίσουν το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα ευάλωτα ε, άτομα και το οποίο περιγράψατε με τόση ακρίβεια και λεπτομέρεια. Θα ήθελα να ξεκάθαρω προς εσάς ότι ε, εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανησυχούμε για αυτήν την κατάσταση και ότι θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε εκ του σύναγκης. Θα πρότεινα επίσης να αποσταλεί η αναφορά προς ενημέρωση στην Επιτροπή Απασχόλησης εκπροσωπώ την Επιτροπή Αναφορών στην Επιτροπή Απασχόληση και πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο. Η Πρόεδρος, ναι, συμφωνώ απολύτως, είναι πολύ σημαντικό και ω μέλος της Επιτροπής Απασχόληση θα ζητήσουμε από εσά να το ε, φροντίσετε αυτό και να την παρουσιάσετε αναλυτικά τον φτάσει. Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο που όρισε σωστά την πολιτική διαμάχη. Θεωρώ πως είναι ειλικρινές να υποθήσει στους αναφέροντες πως βάσει της σα νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αρμοδιότητα βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει πως αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Αλλά το λέω και για τον αναφέροντα πως πρόκειται για μια μακρά διαδικασία. Θα ήθελα να παρακαλέσω όμως και τους αναφέροντες να μην υποχωρήσουν στην Ισπανία να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους εκεί επειδή είναι μια τυπική αντίφαση αφενός θέλουμε να εναρμονίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφετέρου έχουμε την επικουρικότητα δηλαδή αρμοδιότητα των κρατών μελών και στον τομέα αυτό η αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι σαφής Γι' αυτό και θα πάρουμε την μακρά διαδικασία που ανέφερα. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα επίση στην αρμόδια επιτροπή. Γι' αυτό και παρακαλώ του αναφέροντε να μην σταματήσουν, να μην υποχωρήσουν και να συζητούν το θέμα αυτό και περαιτέρω στην Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα ήθελα να απευθυνθώ στι αρχέ της Βαλένθια και να πω πω δεν μπορείτε δεν είστε μόνο εσείς που μπορείτε να στείλετε εκτενείς επιστολές, αλλά και εμείς έχουμε ενδιαφέρουσες μελέτες, τις οποίες θα περιλάβουμε στην απάντησή μας προς εσάς. Θα βρείτε δηλαδή μία μελέτη, την οποία ανάθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ όλους σας για αυτό και θα προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά. Είναι ένας παλιός μας φίλος, Κάτι που ανησυχεί την Επιτροπή είναι η 930 του 2016 σχετικά με την ταχεία κύρωση, υλοποίηση και εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακές. Ο Δαβίτ Χέμερστέιν βρίσκεται εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι, ένας παλιός μας φίλος και πρώην μέλος του Κοινοβουλίου. Έχετε επί πέντε λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο στις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη. Δεν γνωρίζω εάν το Συμβούλιο είναι παρόν εδώ, υπάρχει εκπροσώπηση του Συμβουλίου. Προσκλήθηκαν, αλλά δεν είναι παρόντες. Αυτό είναι απογοητευτικό. Καθώς το Κοινοβούλιο έχει ομόφωνη θέση σχέση με την συνθήκη του Μαρακές. Το, ενώ το Συμβούλιο για τρίτη φορά δεν είναι παρόν ενώπιον της Επιτροπής αυτής. Το πρώτο που θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή είναι να εκφράσει τη λύπη του για την αποσία του Συμβουλίου παρότι προσκλήθηκε για το θέμα αυτό. Όπως είπα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για τις διαπραγματεύσει για τη συνθήκη του Μαρακές. Ο τριμερής διάλογος έχει αρχίσει και παρά την ομόφωνη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρά μια πολύ σαφή αρχική πρόταση, θετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκετά κράτη-μέλη έχουν θέσεις που απέχουν πολύ από αυτές του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απέχουν πολύ από το να οικονοποιήσουν τους στόχους της συνθήκης του Μαρακές για εύκολα προσβάσιμα βιβλία για ανθρώπους με αναπηρίες όρασης. Είχαμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αρμοδιότητα για τη συνθήκη του Μαρακές και σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση των διασυνοριακών ανταλλαγών ρυθμίζεται από το άρθρο 114 της συνθήκης το οποίο είναι αποδεκτό για την Κομισιόν και σύμφωνα με αυτό που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και ενοποιημένου κανόνες για την άρση των περιορισμών του copyright. είναι ακριβώς αυτό που περιέχει η οδηγία για την υλοποίηση της συνθήκης του Μαρακές. Καθίσετε σαφές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κύρωση της συνθήκης. Σημαίνει επίσης πως υπάρχει πως μια διαφοροποιημένη υλοποίηση θα αποτελούσε, αναχώρα θα αποτελούσε παράβαση του 114 θα σημαίνει μια χαοτική υλοποίηση, διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος ιδίως ως προς τα δύο στοιχεία που η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λένε πως πρέπει να ενοποιηθούν, δηλαδή η οικονομική αποζημίωση και η εμπορική διαθεσιμότητα. Παρά τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ομόφωνη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρκετά κράτη-μέλη, πρέπει να αναφέρω κάποια εδώ, η Γερμανία, η Δανία και η Ισπανία ζητούν ακόμα δικαιώματα οικονομικής αποζημίωσης για κάθε βιβλίο. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία θέλουν ο Γερμανικός Οργανισμός Τυφλών να πληρώνει 13 ευρώ και 50 λεπτά για κάθε βιβλίο. Υπόθηκε επίσης που δεν μπορούμε να περιμένουμε τους Αυστριακούς να πλημμυρίσουν την αγορά με έργα για τους τυφλούς. Αυτό θα κατέστρεφε το σύστημα αποζημίωσής μας. Μιλούμε για αποζημιώσεις για απώλειες που δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρξουν, επειδή η συνθήκη του Μαρακές διασφαλίζει αυτό να γίνεται σε μη κερδοσκοπική βάση για τα μέλη των οργανώσεων τυφλών. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί η αιτία της συνθήκης αυτής αφισβητείται βάσει κριτηρίων αγοράς η διάθεση βιβλίων για ανθρώπους με αναπηρίες όρασης δεν θέτει σε κίνδυνο τα κανονικά οικονομικά συμφέροντα κανένας τομέα, ούτε του τομέα των εκδόσεων. Παρομοίως, η Ισπανία υποστήριξε πως ναι, υπάρχει οικονομική αποζημίωση γι' αυτό, αν και επί πολλά χρόνια ποτέ δεν υπήρξε η παραμικρή οικονομική αποζημίωση για βιβλία τα οποία μοιράζονταν με οργανισμούς τυφλούν τυφλών. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώ κάποιε χώρε μιλούν για τέτοια θέματα, αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε που ζητούν κάτι για την εμπορική διαθεσιμότητα. Θέλουν τα πάντα να είναι à la carte. Ότι κάθε χώρα να υλοποιήσει την συνθήκη όπως θέλει. Και αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα και με το γράμμα μιας εναρμονισμένη εσωτερική αγορά όσον αφορά την εμπορική διαθεσιμότητα. Δηλαδή αν το βιβλίο βρίσκεται στην αγορά τότε δεν μπορεί να μοιραστεί εκτός και αν αυτό επιτρέπεται υπό αυτή την νομοθεσία. Η Κομισιόν ζήτησε να μην υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την εμπορική διαθεσιμότητα και την αποζημίωση στα κράτη-μέλη, επειδή το θεωρεί ως εμπόδιο. Η εμπορική διαθεσιμότητα δεν είναι απαραίτητη. Γιατί ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός να έκανε ένα ειδικό αντίγραφο ενός βιβλίου με μεγάλο κόστος, ένα αυτό κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, αυτό δεν θα γινόταν. Το πρόβλημα είναι επίσης το τεράστιο διοικητικό άχθος για βιβλία που κυκλοφορούν κάπου στον κόσμο και σημαίνει επίσης αυξανόμενο κόστος για τον εφοδιασμό των φτωχών και δημιουργεί επίσης νομική αβεβαιότητα. Η εμπορική διαθεσιμότητα και αποζημίωση δημιουργεί αβεβαιότητα όταν υπάρχει διασυνοριακή κοινή χρήση βιβλίων. Έτσι στην Λιθουανία κάποιος θα πρέπει να ξέρει την νομοθεσία των διαφορετικών κρατών μελών για την νομοθεσία και την υλοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση βιβλίων για ανθρώπους με αναπηρίες όρασης. Αυτό που θα ήθελα από την Επιτροπή Αναφορών σήμερα εδώ είναι να ζητήσει από το Συμβούλιο να σεβαστεί το κείμενο στην αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας να σεβαστεί τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανώσεων ανθρώπων με αναπηρίες όρασης ως προς την αιτιολογική σκέψη 11 θα ήθελα η επιστολή αυτή να σταλεί στις ε, αντιπροσωπείες των κρατών μελών και το ΕΒ προκαλεί πολλά προβλήματα ως προς αυτό, αν και η κυβέρνησή του επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταστεί πολύ σαφές πως χρειάζεται μια εναρμονισμένη υλοποίηση της νομοθεσίας αυτής χωρίς εμπόδια και με αυτό το σκοπό η επιστολή αυτή θα πρέπει να αποσταλεί πριν από την επόμενη συνάντηση στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου στις 10 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, David. Νομίζω ότι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα είναι να ζητήσουμε τη Μάργαρετ και τον Πέταρ να τηλεφωνήσουν σε κάποιον πρόσωπο της κυβέρνησης του αφού μας τα λέτε. Αστειευόμουν. Αλλά χρήσιμο θα ήταν εδώ που τα λέμε. Πάντως δεν θέλω να φύγετε από την αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στην, στον κύριο Έβερτ, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον David Hammerstein που έθεσε το θέμα. Θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή, να σας εξηγήσω που βρισκόμαστε από την πλευρά της ε, Επιτροπής, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση της ε, συμφωνίας. Έχουμε υιοθετήσει στις 14 Σεπτεμβρίου της ε, προηγούμενης χρονιάς την πρόταση οδηγίας και κανονισμού. Έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, ο τριμερής διάλογος με τον συνομοθέτη και διαπιστώνουμε ότι το θέμα, στο θέμα αυτό έχει σημειωθεί πρόοδος. Πάντως, τα προβλήματα που ενέφερε και ο κύριος Χάμερστάιν παραμένουν. Η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, δεν συμπεριλάμβανε ε, αυτή την πρόταση για ένα σύστημα ανταποδοτικό και τον έλεγχο με κριτήρια της αγοράς που είναι κάτι το οποίο προήλθε από πρόταση των κρατών μελών. Τα θέματα αυτά είναι βεβαίω ζητήματα συζήτησης με τον συνομοθέτη. Έχουμε διαπιστώσει ότι σημειώνεται πρόοδος και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ανέφερε και ο Σχαμεστάιν επίση το ζήτημα τη κύρωση. Αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στι 14 Φεβρουαρίου του 2017 επικύρωσε, επιβεβαίωσε μάλλον ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην επικύρωση, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος και σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει στο Συμβούλιο την πρόταση αποφάσεως για την επικύρωση. Ε, αυτή η πρόταση αποφάσεως έχει μπλοκαριστεί, αναμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί είχε τεθεί το ζήτημα του κατά πόσον ε, το θέμα αυτό αποτελεί από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Ε, συνολικά και συμπερασματικά θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί το θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Προσπαθούμε να και επιδιώκουμε την ε, επικύρωση της Συμφωνίας του Μαρακές ως το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την Μάργαρετ. Ευχαριστώ τον κ. Χάμερσταν και την Επιτροπή. Στο συγκεκριμένο θέμα έχετε παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο. Το θέμα το συζητάμε στην Επιτροπή από το 2009 και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή έχει, έχουν κάνει σημαντική πρόοδο, έχουν προωθήσει τα πράγματα και είναι λυπηρό να διαπιστώνουμε τι συμβαίνει από την πλευρά του Συμβουλίου και από κορισμένα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την ε, εντολή επικύρωση, ακολουθούσε την ε, πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα αιτήματα των εκπροσώπων των οργανώσεων των τυφλών. και, και, και Στην ε, Δανέζικη Βουλή υπήρξε και μια... Ε, επανήλθε το θέμα σαν να επρόκειτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην είχε, μην είχε λάβει θέση παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει πολλές ψηφοφορίες τις οποίες είχε, είχε, είχε προκριθεί η κύρωση τη συμφωνία του και με μεγάλε πλειοψηφίε. Δεν αντιτάχθηκαν στην καλή πρόταση της Επιτροπής. Στις 16 Μαρτίου ε, οργανώσεις τυφλών διαμαρτυρήθηκαν για τις κολλησιεργία αυτή. Δημιουργούμε λοιπόν προβλήματα ορισμένα κρατημέλη και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε στους διάφορες κυβερνήσεις μας ότι αν καταφέρουμε και δημοσιοποιήσουμε το θέμα, ε, ζήτω που κάηκαν, εάν καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ δεν ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των τυφλών. θέμα είναι το που έχει τεθεί είναι τι θα γίνει με ένα αντίγραφο το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο. Αυτό στην πραγματικότητα θα βοηθήσει την εκδοτική βιομηχανία, δηλαδή την αγορά, εάν το ε, προσβάσιμο αντίτυπο είναι ήδη ε, διαθέσιμο. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το χρονοδιάγραμμα, το χρονικό όριο που ζητάει το Συμβούλιο για να επικυρώσει. Το 2013 υπογράψαμε τη Συμφωνία του Μαρακές και γνώριζαν τα ζητήματα. Και συνεχίζουν να κολλησιεργούν. Αν δεν απατώμε, μάλιστα το 2016 ζήτησε το Συμβούλιο από την Επιτροπή να του υποβάλει και μια πρόταση υλοποίηση τη ε, Συμφωνίας του Μαρακέ. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος, καμία δικαιολογία για όλη αυτή την καθυστέρηση. Έτσι κι αλλιώς μιλούμε και για μια αγορά εξαιρετικά μικρή από οικονομικής απόψεως. Είναι απολύτως ε, παράλογο. Παλαιότερα είχαμε προβλήματα και με τις, με τις γαλλικές ε, αρχές, με την γαλλική κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα. Πιστεύω ότι πρέπει να οργανωθούμε σε πολιτικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Και πέτα, ενημερώστε την κυβέρνηση σας ότι δεν ότι θα τα βρουν σκούρα εάν μάθει ο κόσμος ότι ακολουθούν τις προτάσεις της εκδοτικής βιομηχανίας εις βάρος των τυφλών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να συγκρατήσουμε πως δεν είναι μια ένδοξη σελίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Αυτό που επιβραδύνει την όλη διαδικασία είναι, αυτή η σχέση, αυτό που γίνεται στα παρασκήνια. Δηλαδή είναι ο καυγάς και τις αρμοδιότητες. Σε κανένα δεν αρέσει να εκχωρεί αρμοδιότητες, οπότε τα κράτη-μέλη παρατείνουν τη διαδικασία, προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά εδώ το ζητούμενο είναι οι θυγόμενοι. Και έχουμε 28 κράτη-μέλη και 28 δημόσιες διοικήσεις οι οποίες θα πρέπει να βρουν μια λύση μαζί με την Κομισιόν καθώς η γνώμη του Κοινοβουλίου είναι γνωστή. Η άποψη της Κομισιόν είναι και πολύ κοντά σε αυτήν του Κοινοβουλίου. Τώρα ο καθένας θα έπρεπε να μιλήσει με την κυβέρνησή του. Εκ των έξω δεν έχει νόημα το ότι δεν προχωράει το όλο ζήτημα. Η Κομισιόν με ενθάρρυνε λίγο, διακρίνει κάποια πρόοδο. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, να ασκήσουμε πίεση, σωστά. Το ανοιχτό πνεύμα, επίσης, σωστό. Και σε ποιον μπορούμε να απευθυνθούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει κατά 200% την Επιτροπή Αναφορών και τον αναφέροντα, η Κομισιόν επίσης. Το ρωτημά αγαπητοί Πρόεδρε, είναι πρέπει να γράψουμε μια επιστολή στο Συμβούλιο, να τους πούμε, κοιτάξτε φίλοι, κάντε επιτέλους κάτι και αφήστε τις ιδεολογίες. Επειδή εδώ κρυβόμαστε πίσω από επιχειρήματα, ενώ χρειαζόμαστε ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, την τον καθορισμό των τιμών των βιβλίων, αλλά είναι σαφές πως πρόκειται για μια περιορισμένη αγορά εδώ. Και σε τελική ανάλυση το ζήτημα αφορά ανθρώπους με αναπηρίες. Δηλαδή, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο, επειδή αυτοί παρακολύουν τη διαδικασία. οι Κομισιόν είναι στην πλευρά μας. Γι' αυτό και επιστρέφω το ερώτημα στην Πρόεδρο. Ελενόρα Εύη. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Είναι μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο δημιουργεί την εντύπωση ότι η Ευρώπη ακόμα και για αυτά τα δικαιώματα δεν έχει ενιαία ρύθμιση, ότι υπάρχει κατάτμιση των ρυθμίσεων θα πρέπει ε, να, να δείχνουμε στο συμπέρασμα ότι ενδιαφέρονται περισσότερο τα εμπορικά παρά για, για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν ε, δικαιολογίε. Σα το ξαναλέω και εγώ. Είπαμε τι είναι το Φεβρουάριο του 2017, δεν έγινε τελικά η κύρωση τη ε, συνθήκης. Καθυστέρησε. Είναι απαράδεκτο έχουμε τις σωστές προτάσεις των συναδέλφων και είναι ηθικό μας καθήκον ως Επιτροπής να προσπαθήσουμε και να προστατεύσουμε αυτά τα τόσο θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία συχνά καταπατώνται. Να στείλουμε επιστολή στο Συμβούλιο να τους επισημάνουμε ότι θα πρέπει ε, να διεκπληρώσουν το θέμα ταχύως. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποιος έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση εδώ. Η βαβαρική κυβέρνηση ε, ζήτησε στον Bundesrat να υποστηρίξει να υποστηριχθεί η θέση της όσον αφορά το σύστημα της οικονομική το... οικονομικής ανταπόδοσης. Τρεις φορές. Και μάλιστα ε, συνεχίζουν να το υποστηρίζουν αυτό και στέλνουν ε, mail σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιταλία. Τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο το Ιταλικό εξέφρασαν την υποστήριξή τους, την υποστήριξη τους στην θέση που εκφράζεται και στην αιτιολογική σκέψη 11. Αυτό συμπεριλαμβάνει και μέλη της, Ευρω... της... της κυβέρνησης της Ιταλίας. Παρ' όλα αυτά, η Ιταλική κυβέρνηση στο Συμβούλιο λαμβάνει την αντίθετη θέση. Αναρωτιέται κανείς πώς λειτουργεί η δημοκρατία εδώ χρειάζεται να υπάρξει μια νομική ρύθμιση για να υπάρξει αυτή η εναρμόνιση. Ε, η κατεύθυνση, την κατεύθυνση μας τη δίνει η αιτιολογική σκέψη 11. Εάν δεν ακολουθήσουμε αυτήν θα δημιουργηθεί χάος. Και ξέρετε πού θα καταλήξουμε. Πάλι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το θέλουμε να συμβαίνει αυτό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να φτάνουμε στην κατάσταση τελικά οι δικαστέ του Λουξεμβούργου να επιλύουν τα ζητήματα. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που πολύ έξυπνα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να δώσουμε κατευθύνσεις για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσία. Μιλούμε για θεμελιώδη ε, δικαιώματα και αν η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ξεκάθαρη, δεν θα βασιστούμε, θα, μπορούμε να βασιστούμε στο, θα μπορέσουν να βασιστούν μάλλον οι οργανώσεις τυφλών στο σύμφων, στη, σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ανθρώπων με αναπηρία. για το ζήτημα των εθελοντικών μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων τυφλών και των εκδοτικών, της εκδοτικής βιομηχανίας. Δεν ισχύει ότι η νομοθεσία είναι εναντίον αυτών των συμφωνίων. Δεν υπάρχει τίποτα στην νομοθεσία η οποία να αποκλείει την δυνατότητα μια οργάνωση, μια οργάνωση τυφλών να έχει συμφωνήσει με εκδοτικούς οίκους για να έχει δωρεάν αντίτυπα ή κάτι τέτοιο. Ε, ορισμένες εταιρείες, επιχειρήσεις εκδοτικής βιομηχανίας μας λένε ότι ναι, αλλά αν περάσετε αυτή την νομοθεσία, οι οργανώσεις του ΦΛΟΝ θα πάψουν να συνεργάζονται μαζί μας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Ε, δεκάδες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επικυρώσει ε, τη Συμφωνία του Μαρακές στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία και ο Καναδάς αν δεν απατώμε. Ωστόσο, γνωρίζετε ότι η μεγάλη πλειονότητα των βιβλίων αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ισπανικών, δηλαδή των μεγαλύτερων και πιο διαδεδομένων ε, γλωσσών της, ε, του πλανήτη, εκδίδονται ε, στην Ευρώπη. Η συμφωνία του Μαρακές δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, να έχει ένα ουσιαστικό αντίκτυπο, εάν δεν ε, συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλει η Επιτροπή Αναφορών ε, προ το Συμβούλιο, αποστέλλοντα μια αποστολή ε, υπενθυμίζοντά τους τις υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσει που έχουν αναλάβει με βάση την αιτιολογική σκέψη 11. Η πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Επίσης σα ευχαριστώ για την επιμονή που έχετε δείξει σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι ο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μας είπε ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη η Επιτροπή για την πιθανότητα να καταφέρουμε να υπάρξει συμφωνία. Να σα ενημερώσω επίσης ότι έχει οργανωθεί μια τεχνική ε, συνάντηση. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε και ο, ο, εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Μπορεί να είναι σε αυτή την τεχνική συνάντηση για να προετοιμαστεί. Επομένως σας ζητώ να συνεχίσουμε να έχουμε μια θετική διάθεση επέναντι στα πράγματα αντιλαμβάνομαι τι λέτε, ε, David, ε, να στείλουμε αυτή την επιστολή, όμως θα ήταν περίεργο να σταλεί αυτή η επιστολή ε, και στους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών που είναι υπέρ της ουσιαστικής ε, εφαρμογής της Συμφωνίας του Μαρακές. Πιστεύω θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο αν στέλναμε την επιστολή σε εκείνους που στην πραγματικότητα μπλοκάρουν την επικύρωση. Ο κύριος Χάμεσπεθ. Είναι ξεκάθαρο ότι ορισμένες χώρες έχουν λάβει μια πιο ε, μια επικοδομητική στάση, όπως η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Δανία τώρα που φτάνουμε στην υλοποίηση την πραγματική και η Ισπανία σιγά σιγά αρχίζει να σκληραίνει τη στάση της, η πρόεδρος. Προσωπικά πιστεύω ότι η διατύπωση της επιστολής θα μπορούσε να είναι πολύ αυστηρότερη αν απευθυνθεί μόνο σε εκείνες τις χώρες οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα. Ε, παρά εάν στείλουμε μια επιστολή σε όλους τους μόνιμους αντιπροσώπους. Ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε, να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα και να στείλουμε σε εκείνους. Μάργαρετ, μια μικρή παρατήρηση. Η θέση αυτή είναι η επίσημη θέση του Συμβουλίου. Εγώ συμμετείχα στον προηγούμενο τριμερή διάλογο. Ήταν δύσκολο ο τρόπο με τον οποίο τελικά στο Συμβούλιο συμφώνησε σε αυτή τη θέση αυτή. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να στείλουμε μια επιστολή σε ολόκληρο το Συμβούλιο αλλά δεν είναι μυστικό ποια χώρα δημιουργεί πρόβλημα, το γνωρίζουμε αυτό, ο καθένας από τα εθνικά μας κοινοβούλια. Ε, ε, πιστεύω λοιπόν ότι συνολικά η, θέση της πλειοψηφία του Συμβουλίου είναι αρνητική. Η πρόεδρο. Εντάξει, οκ. Okay. Θα στείλουμε μια επιστολή σε όλους, σε όλους τους μόνιμους αντιπροσώπους στο Συμβούλιο, για να τους δείξουμε ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη τους. Σας ευχαριστώ Μάργαρετ για αυτήν τη διευκρίνηση. Έτσι θα προχωρήσουμε, David. Συνεχίστε τον αγώνα σας και μην τα παρατήσετε. Ο κύριος Χάμερσπιθ, να μείνετε ήσυχοι, Σεσίλια, δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Σε ευχαριστούμε που ήρθες και θα είμαστε σε επαφή. Πάμε τώρα στην επόμενο θέμα που είναι το 16. Είναι η αναφορά 0 986 ε, ναι, του 2015 όσον αφορά το σύστημα προσόντων, κοινωνική αναπηρία, αναπηρία ως προϋπόθεση για εξετάσεις αγωγή. στα πανεπιστήμια. Δεν έχει έρθει ο αναφέρον. Οπότε, με χαρά να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τσόρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. There. Uh, so, indeed... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντως ε, ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με αυτή την ε, αναφορά. Πρώτα-πρώτα, η εκπαίδευση είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητος. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρώτα-πρώτα αντιδράσαμε απαντώντας λέγοντας ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Διότι δεν προβλέπεται το κοινωτικό δίκαιο όσον αφορά αυτή την περίπτωση. Οπότε πρώτα πρώτα έχουμε υπόψη μα την Σύμβαση με των Διαδικαιώματων των Ατόμων με Αναπηρία, το άρθρο 24. Και η Σύμβαση έχει κυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των καλομερών και την Ιταλία. Η Ιταλία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα πρέπει όλοι οι ανάπηροι να έχουν προσβάσει σε αυτές τις εξετάσεις αγωγής και πέραν της συμβάσεως. Να δούμε τι έχουμε ως νομοθεσία, πώς, πώς μπορεί να υπάρξει επέκταση αυτού του δικαιώματος. Έχουμε δηλαδή την ε, οδηγία όσον αφορά την ισότιμη ε, μεταχείριση απασχόληση. Το 2008 αποφασίσαμε να ε, υπάρξει επέκταση του παιδί αυτής της οδηγίας και για την εκπαίδευση και συμφώνησε και το Κοινοβούλιο με, ε, για αυτό το θέμα. Αλλά το θέμα συζητείται στο Συμβούλιο και αυτό σημαίνει ότι λίγα κράτη, κάποια κράτη-μέλη τέλο πάντων δεν ήταν υπέρ αυτής της ε, επέκτασης του ε, για τις οδηγίες για την ισότητα. Να, το πρώτο στοιχείο το οποίο έχουμε. Αυτά είπαμε και στον αναφέροντα και είναι το θεμεμένο σε αυτό και το της σύμβασης του ΙΕ. Τι κάνουμε με αυτήν. Λέμε στα κράτη-μέλη και το έχουν βέβαια υπόψη τους ότι θα πρέπει ε, κάθε τόσο να υποβάλουν κάποιες ε, εκθέσεις στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ. Δηλαδή περίπου κάθε 4 έως 6 χρόνια περίπου. Η Ιταλία πέρσι, τον Ιούνιο δηλαδή του 2016, υπέβαλαν τη σχετική έκθεση για το πώς εφαρμόζουν την σύμβαση και τι κάνουν με τα σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και λίγους μήνες μετά η Επιτροπή του ΟΗΕ απήντησε στην Ιταλία με παρατηρήσεις σχόλια. Και όσον αφορά το άρθρο 24 που αφορά την εκπαίδευση. Και έλεγαν θα πρέπει να του αγκαλιάσει όλους η ρύθμιση. Γιατί υπήρχαν όλοι, ε, κάποια σχόλια επίσης από το μηχανισμό παρακολούθησης ε, της Ιταλίας για την ε, σύμβαση. Υπάρχει εθνικό παρατηρητήριο προς τούτο. Οπότε ε, μία από τις παρατηρήσει που θα μπορούσα να διαβάσω και ας μην εδώ αναφέρω, που είναι η δική μας θέση, είναι ότι η Επιτροπή του ΟΗΕ συστήνει ε, στην Ιταλία ότι θα πρέπει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη ρύθμιση όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και να υπάρχουν σχετικές ε, ε, διευκολύνσεις. Οπότε εδώ έχουμε δύο παράλληλε διαδικασίε που θα μπορούσε να αποσχολήσει τον αναφέροντα. Πρώτα πρώτα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Εθνικό Πρατηρητήριο. Δεν ξέρουμε εάν το έχει κάνει αυτό ο αναφέρον. Και αυτή ε, στο παρατηρητήριο δηλαδή είναι η αρμόδιοι. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν ήδη έχει έρθει σε επαφή ο αναφέρον ε, με το Εθνικό Πρατηρητήριο και αν έχει εξαντλήσει όλα όσα προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία, τότε δικαιούται ο αναφέρον να απευθυνθεί απευθεία ο ίδιο. στην ε, Επιτροπή των Ανθρώπων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Άρα πρώτα-πρώτα εξαντλούνται τα εθνικά ενδικά μέσα και μετά ο ΙΑ. Γι' αυτό ακριβώ και εμεί προτείναμε, συμβουλεύοντα τον αναφέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο. Και τώρα τα μέλη έχουν το λόγο, η Ελεονόρα Εύβοια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εν προκειμένου έχουμε ενωπιόν μας μια κατάσταση κατάφορης ε, δυσμενούς διάκρισης εις βάρος ε, αναπήρων. Και ε, ούτε τώρα μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν μια οδηγία αυτή που αναφέρθηκε η οδηγία δηλαδή κατά της νομής διάκρισης να έχει από το 2008 μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο για άλλη μια φορά γιατί δεν υπάρχει κοινή θέση του Συμβουλίου. Το θέμα είναι το πώς θα εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση. Σε όλες τις πτυχές της ε, απασχόλησης. Μα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κενό στην, κοινωνική, στην νομοθεσία. Τώρα μιλούμε για το πολύ σημαντικό θέμα της εκπαίδευσης. Είναι καταπληκτικό, είναι τρομερό αυτό. Το πρόβλημα για μια φορά είναι το τι κάνουν, τι δεν κάνουν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο παρά τα όσα έχει πει το Κοινοβούλιο. Έχουμε και ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Μαρτίου του 17 όσον αφορά την ισότητα των δύο φίλων στην Ένωση. Και εκεί για πολλωστή φορά τα είπαμε στο Συμβούλιο. Τους είπαμε ότι πρέπει να υιοθετήσουν μια κοινή θέση. Αλλά συνεχώς μας αφήνουν στο περιθώριο, μας αγνοούν. Παρά το ότι συνεχώς τους ζητούμε να ενεργήσουν. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι είναι το πιο σωστό να γίνει. Ε, νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον θα πρέπει να τοποθετηθούμε ως Επιτροπή ίσως αν είναι δυνατόν με κάποια επιστολή όπου θα προβάλλουμε την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε την κατάσταση αυτής της οδηγίας. Να πούμε ότι αυτό που γίνεται ή που δεν γίνεται δεν αποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων. Απευθυνθούμε και στην Ιταλία. Στη χώρα μου, που είναι προκειμένου ο κακός μαθητής. Απευθύνουμε στην Ιταλική κυβέρνηση. Θα τους ζητήσουμε ξεκάθαρα να τοποθετηθούν. Καταπάτηση δικαιωμάτων και κατάφορη ε, δυσμενής διάκρισης για τα θέματα αυτά της εκπαίδευσης. Ναι, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί επειδή στον τομέα της εκπαίδευση ιδίω. η κατάσταση διαμορφώνεται πολύ περίπλοκη. Στη Γερμανία, αν κοιτάξει κανείς, αρμόδια, συναρμόδια για την εκπαίδευση είναι τα ομόσπονα κρατήδια σε αντιστοιχεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι η Επιτροπή Αναφόρων ίσω ίσως οι αρμοδιότητες της να μην αρκούν. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιες, όλες οι αρμόδιες επιτροπές με αυτό. Έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο της υπερβολικής ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο της μεταφοράς σε εθνικό δίκαιο, πρέπει στα σχολεία πρέπει να μπουν ασανσέρ ανελκυστήρες για παιδιά με αναπηρίες, αλλά τώρα έχουμε περισσότερους ανελκυστήρες από παιδιά με αναπηρίες. Δηλαδή βάλαμε ανελκυστήρες σε κτίρια, τους οποίους δεν χρειάζεται κανείς. Αυτό είναι γερμανική νομοθεσία, όχι ευρωπαϊκή. Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά, δηλαδή έχουμε ανελκυστήρα που δεν χρησιμοποιεί κανένα εδώ και 10 χρόνια, τότε όλοι υποδεικνύουν τι Βρυξέλλε. Γι' αυτό και θα παρακαλούσα η συζήτηση να γίνει με, επί μια βάσης. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ περιπλοκός τομέα και θα ήθελα η Ειδική Επιτροπή να ασχοληθεί, η Αρμόδια Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα. Ευρωπαϊκή Εναρμόνιση είναι πάντα καλά, κάτι καλό, αλλά λαμβάνοντα υπόψη τι περιφερειακέ ιδιαιτερότητε. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό ζούμε. Και πρέπει να βρούμε μια ρύθμιση η οποία να είναι ικανή για την πράξη. Ίσως η όλη αυτή καθυστέρηση να οφείλεται στο ότι δεν τολμούμε να προσεγγίσουμε το θέμα ως Κομισιόν μπορούμε να πούμε επίσης το εξής, αγαπητά κράτη-μέλη, εάν δεν θέλετε να αρχίσετε επικοδομητικές συζητήσεις, τότε θα πρέπει την οδηγία να την κάνουμε κανονισμό. Επειδή το καλό που έχουν οι οδηγίες είναι πως έχει περιθώρια υλοποίηση στα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να, όλη αυτή την ιστορία να την κάνουμε ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Σε 15 λεπτά είναι πολύ δύσκολο να τελειώσουμε με το θέμα. Υπάρχει μια σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, με την οδηγία κατά των διακρίσεων. Θα μπορούσε να υποθεί πως ακόμα βρίσκεται υπό απεξεργασία, υπό συζήτηση στο Συμβουλίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει εμπλακεί στο Συμβούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μια επιστολή, όπως πρότεινε η Ελεονόρα στην Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας της να απεμπλέξει την κατάσταση όσον αφορά την οδηγία αυτή. Αυτό θα ήταν το ένα. όπως σωστά τόνισε η Κομισιόν, δεν μπορεί να παρέμβει στην παρούσα περίπτωση, καθώς δεν υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μία επιστολή στον αναφέροντα και να τον προσκαλέσουμε, να τον προτρέψουμε να καταθέσει την, την περίπτωση στο Εθνικό Παρατηρητήριο που βοηθά θύματα διακρίσεων και παρακολουθεί την υλοποίηση των ευρωπαϊκών συνθήκων ή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε και στη συνέχεια να στείλουμε την αναφορά επειδή είναι ξεκάθαρα εθνική αρμοδιότητα, αλλά μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στους Ιταλούς ζητώντας τους να απεμπλέξουν την κατάσταση και να ενθαρρύνουμε τον αναφέροντα να απευθυνθεί στο Εθνικό Παρατηρητήριο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τέλεια. Τώρα έχουμε μια πολύ ασυνήθιστη κατάσταση στην Επιτροπή αυτή. Έχουμε 25 λεπτά μέχρι να έρθει ο Φραντ Τίμερμαν, ο πρώτο αντιπρόεδρο τη Επιτροπής, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να βγείτε, να ξεκουραστείτε, αλλά να ξανάρθετε στι 11 παρα 5, επειδή είναι Ολλανδό και είναι πολύ στην ώρα του. Θα είναι εδώ στις 11 παρα 5 και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν όλοι καθόμασταν Πολύ ωραία στις 11. Εντάξει. Απολαύστε το διάλειμμα σας και Γιάρεκ έχεις 20 λεπτά για να πιεις έναν καφέ ή για να πάρεις τηλέφωνο. colleagues and friends, dear Vice President Timmermans, it's... Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, κύριε Αντιπρόεδρε Timmermans, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Αναφορών. Είναι τιμή για εμένα να σας καλωσορίζω στην αγαπημένη σας Επιτροπή, ελπίζω. Στο πλαίσιο το ετήσιο του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Επιτροπών του Κοινοβουλίου Ήδη από την περσινή χρονιά το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης ήταν πολύ θετικό και ελπιστούμε ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Έχουμε το πρόγραμμα εργασιών του 2017, την υλοποίηση του φετινού προγράμματος της Επιτροπής και την προετοιμασία για το πρόγραμμα εργασιών για το 2018. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε σήμερα. Μετά την ανταλλαγή μου και τον κύριο Τίμερμαν θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα αποστείλουμε και στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών και θα αποτελέσουν μέρος της, του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα προσθέσω τίποτα παραπάνω. Δίνω κατευθείαν το λόγο στον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν. Σας ευχαριστώ. Ε, είμαι ιδιαίτερος που απευθύνομαι στην Επιτροπή σα για άλλη μια φορά. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω για να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Η επιθυμία μου είναι να συζητήσω μαζί σας, γιατί η Επιτροπή σας βρίσκεται πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη από οποιαδήποτε άλλη, γιατί εσείς βρίσκεστε σε άμεση επαφή με τους πολίτες, με τις αναφορές που λαμβάνετε από αυτούς και αν κανείς εξετάσει τα διάφορα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους πολίτες και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και αυτό είναι φυσικά το Brexit. Γιατί θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τα δικαιώματα των πολιτών με διάφορες μορφές και πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μας να ακολουθήσουμε τον όρκο του Ιπποκράτη, να μην προξενήσουμε βλάβη. Αυτή να είναι στο δυνατόν πιο περιορισμένη όσον αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι η άποψή μου και είναι και πιστεύω και ότι η κατεύθυνση προς την οποία μας πηγαίνει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, το οποίο μας ζητά να ξεκινήσουμε την όποια διαπραγμάτευση με γνώμονα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και πιστεύω ότι αυτό μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαριστεί και με τις κατευθυντήριες οδηγίες διαπραγμάτευσης που θα υιοθετήσει το Συμβούλιο. Ε, και ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί και από τη δικιά του την πλευρά για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχει κάτι που δεν άλλαξε από την προηγούμενη μας συνάντηση. Και αυτό είναι η πεποίθησή μου ότι ε, το έργο της Επιτροπής σας είναι εξαιρετικά σημαντικό, το παρακολουθώ από πολύ, πολύ στενά και το επιβεβαιώνω, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα. Από την προηγούμενη μας συνάντηση έστειλα επιστολή στον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Ολλανδία ζητώντας οι διάφορες αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες να την χάνουν ε, επεξεργασίας και να στέλνουν τις απαντήσεις. Γιατί συχνά χρειάζεται συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και κρατών μελών. Συχνά στο εθνικό επίπεδο, αλλά πολλές φορές επίσης και στο περιφερειακό από την πλευρά μα, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποτεδήποτε η Επιτροπή Αναφορών μα ζητάει πληροφορίε, προσπαθούμε να σα τι αποστέλνουμε χωρί κολυσιεργία, χωρί να καθυστερούμε. Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που σα ανησυχεί και έχω ζητήσει από του συναδέλφου μου να φροντίζουν να τηρούνται οι προθεσμίε. Ε, όλες οι αναφορές που μας αποστήλατε κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2016 μπορώ να σας πω ότι καταφέραμε να απαντήσουμε σε όλες εντός τριών μηνών και στο 75% των ε, αναφορών καταφέραμε η απάντηση να έρθει σε δύο μήνες ή ακόμα και ε, πιο σύντομα. Μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά τουλάχιστον ε, θα έλεγα ότι έχουμε σημειώσει μια κάποια πρόοδο εδώ. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία μας από τώρα μέχρι το τέλος των θητιών της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή συνεργασία που καταφέραμε να χτίσουμε τα πρώτα χρόνια. Βεβαίως, αν εντοπίζετε εσείς κάποιους τομείς στους οποίους θα ε, πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθούμε και ότι δεν ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις σας, ε, μπορείτε να μου τους αναφέρετε, να το συζητήσουμε. Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα στο οποίο συζητούμε πάντοτε, κάθε φορά που συναντιόμαστε, είναι η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Ε, συζητιέται πολύ, όπως γνωρίζετε, το πόσο απομακρυσμένοι είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί από τους πολίτες και πιστεύω ότι είναι χρέος όλων μας να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών την προσπάθεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να τους δείξουμε ότι αυτό είναι που χρειάζεται για να ευημερούμε και για να είμαστε περισσότερο ασφαλείς στο μέλλον. Ε, Μέσω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τη συμμετοχική δημοκρατία δημιουργώντας αυτή την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Από το 2012 έχουμε 50 πρωτοβουλίες εγγραφή που καλύπτουν πολλά και διάφορα θέματα. Αλλά να είμαι ξεκάθαρος δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ε, και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε οποιαδήποτε ε, λύση, οποιοδήποτε βήμα που θα το βελτιώσει είναι στο τραπέζι. Τους επόμενους μήνες θα κάνουμε προτάσεις ε, για τροποποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά τις εγγραφές ε, πρωτοβουλειών, της διαδικασίας για να εγγραφεί μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας, έχει ζητήσει να το πράξουμε αυτό πολλές φορές. Έχω εξετάσει προσεκτικά τι ιδέε που έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών για να παίζει το ρόλο που τη αναλογεί. Η Επιτροπή του επόμενου μήνες θα καταθέσει πρόταση ε, τροποποίησης του κανονισμού που αφορά στην πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών θα είναι περίπου την ίδια περίοδο που γίνεται και η εκφώνηση του λόγου του State of the Union από τον Πρόεδρο αυτό βεβαίως, ε, σε αυτό βεβαίως θα ήμουν ιδιαίτερος ευτυχής αν μου κάνετε κάποιο σχόλιο, κάποια πρόταση για να την λάβουμε υπόψη μας. κλείνοντας. Οι αναφορές είναι ένας τρόπος να έρθει κανείς σε επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά γνωρίζετε ότι οι πολίτες έχουν πολλούς τρόπους για να εκφράζουν τις απόψεις τους. Αν κάποιο θέλει να συγχαρεί έναν τραγουδιστή που πιστεύει ότι είναι καλό, μπορεί να το κάνει από τον καναπέ του σήμερα. Ε, εύκολα. Ενώ στι δημοκρατικέ διαδικασίε που έχουμε, οι πολίτε ερωτούνται και φράζουν τι απόψει του μόνο μια φορά στα τέσσερα χρόνια. Άρα δεν ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες περιμένουν από εμά και αναμένουν να συμμετέχουν στα κοινά. Δεν λειτουργεί πια το παλιό σύστημα δώσε μου την ψήφο σου και επί τέσσερα χρόνια θα σε εκπρόσωπο και εντάξει. Ε, όταν μια πρωτοβουλία έρχεται από την επιπλευρά τη Επιτροπή, συζητιέται ένα θέμα εδώ, οι πολίτε απαιτούν να το γνωρίζουν. Ε, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών, πιστεύουμε ότι η, χρήση, η μεγαλύτερη χρήση του ίντερνετ για τη δημόσια διαβούλευση είναι και αυτό ένα βήμα προς το μέλλον, μια κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε. Ε, σταματώ σε αυτά και ευχαριστώ να ακούσω για τις δικές σας παρατηρήσεις. Η Πρόεδρος. Είναι πολύ ευχάριστο ε, το, η πρότασή σας για τροποποίηση του κανονισμού για την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών θα έρθει ε, ήδη φέτος. Θα ξεκινήσουμε από τους συντονιστές ε, την ανταλλαγή των απόψεων και μετά στα υπόλοιπα, θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη. Ξεκινώ με τον Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς Πιστεύω πως ο επικοδομητικός διάλογος με τους επιτροπές είναι μια θαυμάσια ιδέα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για το ότι εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία και προσωπικά στην Επιτροπή Αναφορών. Το ζητούμενο δεν είναι ανά πέντε χρόνια να ρωτούμε τους πολίτες μέσω των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μεταξύ των εκλογών και εκεί αποφασίζεται και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι καλό ή όχι και η Επιτροπή Αναφορών. Εμείς θεωρούμε πως είμαστε ένας μηχανισμός διαλόγου. Είμαστε κοντά στον πολίτη. και είμαστε το κοιτίο παραπώνων των πολιτών. Δεύτερη γενική παρατήρηση, η συνεργασία με την Κομισιόν έχει βελτιωθεί, μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, είναι σαφές αυτό, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως έχουμε κάνει ένα καλό βήμα βήμα μπροστά. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουμε ακόμα κάποιες επιφυλάξεις. Θα θέλαμε μια πιο στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, επίσης όσον αφορά γνωμοδοτήσεις και τοποθετήσεις στην Επιτροπή Αναφορών. Η Κομισιόν όμως είναι πάντα εκεί, πάντα δίνει απαντήσεις. Τρεις σύντομες ερωτήσεις όμως. Η πρώτη για το Brexit, το είπατε στην εισαγωγή σας. Έχουμε φυσικά δύο ομάδες στην Επιτροπή Αναφορών. Έχουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά φυσικά έχουμε και Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι ζουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε κάποιες λύσεις, προσεγγίσεις για λύσεις για τις δύο ομάδες αυτές. Τι έχετε σκεπτεί σχετικά με αυτό. Ενδιαφέρον έχει επίσης πως Βρετανοί πολίτες απευθύνονται σε μας και μας λένε παρακαλούμε βοηθήστε μας όταν έρθει το Brexit. Πιστεύω πως αυτό είναι θετικό επειδή μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις, σχέσεις για μετά το Brexit. Δεύτερη ερώτηση, εντελώς άλλο θέμα, προστασία μειονοτήτων. Στις νέες χώρες, στα νέα κράτη-μέλη, έχουμε μέρει το φαινόμενο της διασφάλισης της προστασίας των μειονοτήτων, που εξαρτάται επίσης από το ποσοστιαίο μερίδιο τους επί του πληθυσμού. Εάν έχω χ επί του πληθυσμού, τότε αποκτώ το δικαίωμα δίγλωσης επεξεργασίας στη δημόσια διοίκηση, δίγλωσσων πινακίδων κυκλοφορίας. Στη Γερμανία αυτό που έχει γίνει πολλές φορές σε περιπτώσεις είναι μια διοικητική μεταρρύθμιση των διοικητικών περιφερειών με αποτέλεσμα στατιστικά να εξαλείφονται οι μειονότητες. Ο αριθμός τους, ο απόλυτος αριθμός παραμένει ο ίδιος, αλλά ο σχετικός αριθμός χάνεται. περιπτώσεις που έχουν φτάσει στο συνεργατικό δικαστήριο έχουν απορριφθεί λόγω περίεργης επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης. Θα ήθελα να ρωτήσω, εμείς εδώ έχουμε δυνατότητα να παρέμβουμε, να προστατεύσουμε τις μειονότητες όταν έχουμε στατιστικά τεχνάσματα. Το ακούσαμε όχι μόνο από την Πολωνία, αλλά και από άλλες νέα κράτη-μέλη. Τρίτη ερώτηση, πάλι εντελώς άλλο θέμα. Το ψήφισμα για την ενδεξία των παιδιών. Τον Απρίλιο του 2016 είχαμε ένα πολύ ωραίο ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημείωσα τρία πράγματα για τα οποία ζητήσαμε από την Κομισιόν να λάβει μέτρα. Θέλαμε έναν ευρωπαϊκό αριθμό εκτάκτου ανάγκης για την περίπτωση κακοποίησης παιδιών. Επίσης θέλαμε θέσεις εκπαίδευσης για κοινωνικούς λειτουργούς που θα ασχολούνται με διασυνοριακές περιπτώσεις ή θα ξέρουν πώς αντιμετωπίζονται και τρίτο και σημαντικότερο θέλαμε να ζητήσουμε από την Κομισιό να καταρτήσει κατευθυντήριες γραμμές για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεσμικά μέτρα προστασία των παιδιών που έχουμε, καθώ έχουμε διαπιστώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πω το κύριο πρόβλημα σε τέτοιε περιπτώσει είναι πάντα η άγνοια. Ο πολίτης δηλαδή δεν γνωρίζει το σύστημα του άλλου κράτους μέλους. Οπότε είπαμε πως χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων προς όφελος των παιδιών. Η Κομισιόν βρίσκεται από την πλευρά μας με τις καλές μας ιδέες. Πώς το, πώς το βλέπετε. Θα συμβεί κάτι στο όρατο μέλλον. Το ψήφισμα το ψηφίσαμε το 2016 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από μια μακρά διαδικασία στην Επιτροπή Αναφορών. Γι' αυτό και η ερώτησή μου υπάρχει κάτι από πλευρά σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστέ δεν είναι παρόντες. Το λόγο έχει ο κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, I will speak for the ECR for myself. That's for obvious. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του ΣΥΑΡ για την ε, συμμετοχή σας στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι βοηθάει η παρουσία σας ε, για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία της Επιτροπής Αναφορών με την ε, Κομισιόν. απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι μέσα από τη διαδικασία των αναφορών αποδεικνύεται πάρα πολλές φορές ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρανομούν. Και επομένως θα πρέπει να αξιοποιεί την ευκαιρία η Κομισιόν θέματα που βγαίνουν εδώ από την Επιτροπή Αναφορών να αποτελούν και αντικείμενο ενός ντοσιέ της Κομισιόν προκειμένου να παραπέμπονται τα κράτη-μέλη τα οποία ε, παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα επανέλθω σε δύο θέματα τα οποία τα έχουμε ξανασυζητήσει. Το πρώτο αφορά την εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα. Το μνημόνια είναι συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ της Τρόικας και της Ελλάδας και πολλές διατάξεις παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζουν τον χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τέτοιες αναφορές εδώ σε πολλά θέματα που έχουν έρθει και θα έρθουν και την, τον επόμενο μήνα μια σημαντική αναφορά του δικηγορικού συλλόγου του Αιγείου για τα θέματα αυτά. Οι απαντήσεις που παίρνουμε από την Κομισιόν είναι ότι ξέρετε κάτι, είναι ελληνική νομοθεσία που εφαρμόζεται, επομένως δεν έχει να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο παρατηρήσεις αυτό γιατί μου αρέσει ο διάλογος μαζί σας να τον συνεχίσουμε στο θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα το μνημόνιο, το Memorandum of Understanding υπογράφεται από την Κομισιόν και τους υπόλοιπους της Τρόικας με την Ελλάδα. Άρα έχει γνώση η Κομισιόν του τι θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Δεύτερο θέμα και πιο σημαντικό η ελληνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται κατ' εντολή και επιταγή των δανειστών παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί λοιπόν, εφόσον έχουμε τεκμηριωμένη παραβίαση των, του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι στο δικαίωμα της περιουσίας, όταν μειώνει τις συντάξεις Φερρυπίν, παραβιάζεται το δικαίωμα της περιουσίας, τότε η Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό όπως αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα. Δηλαδή αν έχουμε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει τότε να παραπεμφθεί το κράτος το οποίο παραβιάζει την νομοθεσία. Βέβαια εδώ δημιουργείται μια αντίφαση. Πώς θα παραπέμψει η Κομισιόν την Ελλάδα για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου όταν η ίδια Κομισιόν ως μέλος της Τρόικας επιβάλλει στην Ελλάδα να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία. Νομίζω αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα. Είναι αυτή η αντίφαση, η σύγκρουση συμφερόντων Τη ίδια τη Κομισιόν. Η Κομισιόν θα είναι Κομισιόν, θα είναι ο The Guardian of the Treaties ή θα είναι εκπρόσωπο των δανειστών. Αν δεν λυθεί αυτή η αντίφαση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και το δεύτερο θέμα και πολύ σύντομα έχει να κάνει με τις μετεγκαταστάσεις των προσφύγων από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές στο ζήτημα αυτό. Έχουμε τους ίδιους τους κατοίκους των νησιών οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα σήμερα στα νησιά του Αιγαίου, δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση. Υπάρχει συμφωνία για 160.000 μετεγκαταστάσεις από Ελλάδα και Ιταλία σε άλλες χώρες. Όμως, πριν μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, η Κομισιόν και νομίζω ο κύριος Αβραμόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν 160.000 μετεγκαταστάσεις από Ελλάδα και Ιταλία, αλλά μόνο 33.000. Δηλαδή, θα μειωθούν οι μετεγκαταστάσεις κατά 75% που σημαίνει ότι από την Ελλάδα δεν θα φύγουν 66.400 αλλά γύρω στις 16.000. Επομένως αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να συνεχιστεί και θέλω να ξέρω θα ισχύσει αυτό. Αν ισχύσει αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην Ελλάδα γιατί έχουμε χιλιάδες πρόσφυγες και κυρίως έχουμε χιλιάδες παράνομους μετανα... μετανάστες. Και δεύτερον, θα παραπέμψετε τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν την αρχή της μετεγκατάστασης. Θα τα πάτε στο δικαστήριο. Γιατί άκουσα τον κύριο Αβραμόπουλο που είπε ότι δεν θα γίνουν παραπομπές στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αν παραβιάζετε το δίκαιο της Ένωσης δεν πρέπει να έχουμε μέτρα. Άλλωστε και εσείς ο ίδιος σε κάποια ολομέλεια της Ευρωβουλής που συζητήσαμε το θέμα είπατε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τίμερμαν, για το ότι ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Το 2014 αναλάβατε καθήκοντα. Τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πως οι υποθέσεις των πολιτών θα βρεθούν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και θα γίνουν η μεγαλύτερη μας πρόκληση, ιδίως σε σχέση με το Brexit. Θα πρέπει να διακρίνουμε πως η εκπροσώπηση του, των συμφερόντων των πολιτών είναι το σημαντικότερο. Η Επιτροπή μας αποτελεί μια διαρκή σύνδεση με τους πολίτες, επειδή εδώ μπορούν να καταγγείλουν πράγματα, εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να καταγγελθεί, και μπορούν να βασιστούν στο ότι θα τους εκπροσωπήσουμε αντίστοιχα. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, ένα χρόνο μετά την τελευταία φορά που ήρθατε στην Επιτροπή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με ένα θέμα που μας ανησυχεί πολύ, όπως και εσάς, όπως είπατε, την αναθεώρηση του άρθρου 51 για αναφορές, αιτήματα ποια είναι η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών που κατοχυρώνονται από τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα έχουμε μια πολύ περιοριστική ερμηνεία. Και τι λέτε για την άποψη της Επιτροπού Γιούροβα, η οποία είπε πως ανησυχεί επίσης σχετικά με αυτό. Από ό,τι φαίνεται έχουμε σχετικές συζητήσεις, έχουν προχωρήσει. Και ποιες είναι οι προσδοκίες σας ή με ποιο, ποιο σχέδιο δράση μπορούμε να περιμένουμε. Επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε πως όλα τα αφιστάμενα εργαλεία θα είναι σκόπιμα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν σκοπό να λύνουν τα προβλήματα των πολιτών. Το άρθρο αυτό δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το γρηγορότερο δυνατόν. Επειδή βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία, στην οποία είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα επίσης να θίξω ένα άλλο θέμα. Σας είχαμε θέσει το ίδιο ερώτημα και πέρυσι. Τι γίνεται με την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές. Η αποφασιστικότητα της Κομισιόν στο θέμα αυτό είναι σαφώς ορατή. Άσκησε πίεση να προχωρήσει το ζήτημα. αλλά πρέπει να υποθεί πως το ζήτημα αφορά 30 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και το Συμβούλιο προφανώς εδώ δεν επιδεικνύει συνέπεια. Ποια είναι η θέση σας σχετικά με αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών. Μπορούμε να συμβάλλουμε με κάποιον τρόπο. Τι μπορούμε να κάνουμε στις χώρες μας, απέναντι στις κυβερνήσεις μας και τους πολιτικούς μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μία ερώτηση ακόμα που θα ήθελα να θέσω, που σχετίζεται επίσης με τα πολιτικά δικαιώματα και την υποχρέωση της Κομισιόν να επιβλέπει την εφαρμογή των συνθήκων. Σκέπτομαι την κατάσταση στην Ουγγαρία, όπου τα θε, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει υποχωρήσει αισθητά. Απευθύναμε ήδη την περασμένη εβδομάδα μια ερώτηση σε εσά και απαντήσατε πως όσον αφορά τις νέες τροποποιήσεις μιας νομοθεσίας στην Ουγγαρία, η Κομισιόν είχε ήδη τοποθετηθεί. Εδώ το 2012 είχε μπει μία αναφορά και η Κομισιόν είχε ήδη δραστηριοποιηθεί. Αναφέρομαι στο νόμο για την πανεπιστημιακή παιδεία. Και είπαμε ότι υπάρχει εδώ θέμα δικαιωμάτων των Ουγγρών πολιτών μεταξύ άλλων διότι είπαμε ότι αυτό αφορά παραβίαση της πνευστημικής ελευθερίας και κατέβηκε ο κόσμος στο πεζοδρόμιο δεκάδες χιλιάδων ζητήθηκε αλληλεγγύη και να αναλάβει πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποκλείεται το να ξεκίνησε κάποια διαδικασία κατά τη Ουγγρική κυβέρνηση και να υπάρξει κάποιο σοβαρό διάλογο. Μπορείτε να μα πείτε τι είδου διάλογο θα γίνει και πόσο σοβαρό αυτό θα είναι. Συνάδελφοι, όλοι μιλάτε πολύ, επί πολλή ώρα, άρα λιγότεροι θα έχουν ώρα για να μιλήσουν. Οπότε περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο. Κυρία Ροζιέρη, έχετε το λόγο. Κάτι λέει η κυρία Άουκεν, αλλά μικροφώνου. Μην μιλάτε μεταξύ σας, λέει ο Πρόεδρος, να ακούσουμε την κυρία Ροζιέρ. Ε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα. Και έτσι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. να συζητήσουμε για το Brexit αλλά έχουμε τώρα και την δεξιά που πέρασε στο δεύτερο γύρο των εκλογών στην ε, Γαλλία. Πολύ σημαντικό. Να το λάβουμε υπόψη. Ε, επίσης να λάβουμε υπόψη την πολιτική συγκυρία σε όλη την Ευρώπη. να λάβουμε υπόψη το ότι ο κόσμος θέλει να είμαστε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι προτάσεις σας αναμένονται επομένως με αγωνία. Έτσι θα έρθουμε κοντά στους πολίτες. Και σε σχέση με αυτό, για πέστε, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της ε, Ένωσης. Μας μίλησατε για διαβούλευση εσείς. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για το πώς το βλέπετε υπάρχουν κάποια προβλήματα σήμερα, πώς μπορούμε να προσθέσουμε την διαδικασία για την σύλλογη των υπογραφών όσον αφορά την εμπλοκή των πολιτών. Είναι ένας τομέας που θα ήθελα να μου πείτε. Τι γίνεται με το EU Pilot. Εμάς εδώ στην Επιτροπή Αναφορών θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, δυσλειτουργίες Υπάρχει και διαδικασία επί παραβιάση, η παραβάση του γενετικού δικαίου που θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η δυνατότητα ε, προσφυγής. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή Αναφόρων. Πώς θα συνδέσουμε την διαδικασία pilot με τις παραβάσεις αυτές. κάτι άλλο το να ληφθεί υπόψη αυτό που θέλουν οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους. Είχατε ξεκινήσει μια διαβούλευση και το Κοινοβούλιο επίσης με μεγάλη πλειοψηφία το είχε ζητήσει αλλά δεν έκανε τίποτα η Επιτροπή. Να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία και μιλώ για τις γεωγραφικές ενδείξεις των γεωργικών προϊόντων. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, τα ζητήσαμε. Δεν είναι βέβαια θέμα στενά αναφορών, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε. Σας άκουσα και μας είπατε ότι πιέσατε τις κυβερνήσεις να δίνουν απαντήσεις. Πολλές φορές όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο όσον αφορά τις αναφορές. Ή δεν λένε τίποτα ή αργούν ή τέλος πάντων οι απαντήσεις που δίνουν είναι ανεπαρκείς. Άρα παρακαλώ να το ξανακάνετε, να τους πιέσετε να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών. Από την άλλη μεριά και η Επιτροπή πολλές φορές δίνει ανεπαρκείς απαντήσεις. Δεν αγγίζουν οι απαντήσεις αυτά που θέλουν οι αναφέροντες. Εμείς είμαστε σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Νομίζω ότι και εσείς θα πρέπει να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια. Να υπάρχουν αυθεντικές απαντήσεις γιατί έχουμε παραβιάσει ας πούμε οδηγιών από κάποιο κράτος. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, κυρώσεις γιατί ε, αν δεν υπάρχει κύρωση τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν το ίδιο τροπάρι και ο κόσμος θα συνεχίσει να εφίσταται τις συνέπειες αυτής της τακτικής, να εφίσταται την αδικία. Είναι καλά μαντάκτα για αυτόν τον κανονισμό που αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών και είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί τώρα έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και γερό Είπαμε ότι έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν παγώσει 3 εκατομμύρια για το TTIP, 1 εκατομμύριο για ε, το κοινόχρηστο νερό. Ε, σίγουρα και αυτές οι εξελίξεις επιδρούν πάνω σε αυτό το φαινόμενο της απομάκρυσης του κόσμου. Ακριβώς δεν θα πρέπει μόνο στις εκλογές να ασχολούμαστε με τον κόσμο. Α, ήδη έχουμε τώρα το Brexit. Τι θα γίνει άμα κι άλλη χώρα κάνει δημοψήφισμα. Θα βρεθούμε ενώπιον και άλλες έκπληξεις. Έχουμε βέβαια σαν συνέπεια όλων αυτών και την άνοδο της ακροδεξιάς. Ακριβώς γιατί ο κόσμος υποφέρει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, τέλος τη γνώμη της Επιτροπής και για το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Γιατί οι διεθνείς παρατηρητές δεν συμφωνούν για τα όσα πρόκειται να γίνουν, για όσα, όσα συνέβησαν. Με το Ισραήλ έχουμε προτιμησιακή συμφωνία. Στο άρθρο 2 λέει ότι εάν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ανασταλεί η συμφωνία. Αλλά βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα στην Παλαιστίνη. Είναι περίπλοκη η πολιτική, όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάνω απ' όλα. Θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρα. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία, είδατε τι έγινε και στην Ολλανδία. Στο Τσακ γλιτώσαμε από την ακροδεξία. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξουν στην κοινωνία. Επομένως να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την απομάκρυνση των πολιτών από την Ένωση. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Ο αγαπημένος μου εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ θα πρέπει να σταθώ σε ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό για να αποκαταστήσουμε ή μάλλον να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες. Και αυτό είναι η χρηστή δίκηση. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηστή δίκηση. Δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια, το ξέρετε. Είναι γνωστό το πρόβλημα στο Συμβούλιο, ότι είναι απολύτως ε, αδιαφανές. Εντάξει, δεν γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά στους βαθμό που μπορείτε, μπορείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσετε για τη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική για τους πολίτες για να μπορούν να παρακολουθούν τι συμβαίνει και για να, και για να προστατεύει λοιπόν τους πολίτες αλλά και να προστατεύει αν θέλετε τους υπαλλήλους, την δημόσια διοίκηση γιατί έτσι μπορούμε να προσελκύουμε και καλύτερους υπαλλήλους. Και έρχομαι στο ζήτημα το μεγάλο των συγκρούσεων συμφερόντων. Όταν δηλαδή έχουμε μια αρχή η οποία λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματος των πολιτών, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν αρκεί απλώς να δηλώνει κανείς ότι δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων και μετά να πρέπει να γίνει μια εξέταση να δούμε αν μήπως υπήρχε ε, ιδιαίτερα στο ζήτημα των σχέσεων με επιχειρήσεις, με βιομηχανίες, με συμφέροντα τέτοιου χαρακτήρα. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί. Γνωρίζω ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά σε πολύ υψηλό επίπεδο, που, οι οποίοι ακριβώς πριν λάβουν υψηλή θέση στην Κομισιόν ήταν λόμπιστοι, ήταν ε, ε, εκπρόσωποι επιχειρήσεων που μάλιστα στον ίδιο τομέα δραστηριοποιούνται και αμέσως μετά βρέθηκαν στην Επιτροπή. Αυτό πως μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Μπορεί να είναι εξαιρετικό ε, εν λόγω εργαζόμενος βάλλος αλλά ε, πώς διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες για αυτό. Πρέπει να μην υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων για να υπάρχει εμπιστοσύνη και αυτό είναι ξεκάθαρο σε, όλους τους, ε, σε όλα τα επίπεδα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης γιατί όλα αυτά λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν και επηρεάζουν τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε Επίτροπε που ήρθατε. Στη συνέχεια των όσων είπε η κυρία Άουγκεν, θέλω κάτι να σας ζητήσω, να σας ρωτήσω τι γίνεται με τη σύγκρουση συμφερόντων, το revolving doors. Επανειλημμένα το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι υπάρχουν κενά στη ρύθμιση. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Τι γίνεται με τους ε, ε, υπαλλήλους που φεύγουν από την Κομισιόν και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο γίνεται και στις περιφερειακές υπηρεσίες της κοινότητας. Έγινε κάποια έρευνα πρόσφατα στην Ιταλία και αποκαλύφθηκε το μέγεθος του προβλήματος. Δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την επαγρύπνηση για τα φάρμακα και η Transparency International πριν από λίγες ε, εβδομάδες έφερε στο φως το ότι περίπου το 30% των ευρωβουλευτών και 50% των επιτρόπων φεύγουν από την πολιτική πάνε και δουλεύουν σε κάποιες ε, οργανώσεις, σε κάποια γραφεία λόμπι. Ε, έτσι κι αλλιώς εκούσια είναι η ρύθμιση για αυτό το μητρό. Έχουμε όλους αυτούς τους περιορισμούς όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας. Αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί και ρυθμίσεις για το τι γίνεται μετά τη θητεία. Και έχουμε το άρθρο 245 που ακριβώς αφορά το τι θα πρέπει να κάνουν οι επίτροποι κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Μιλά για την υποχρέωση εντυμότητα, μιλά για κάποια πλέον εκτήματα κλπ. Επίσης έχουμε αυτό το cooling off των 18 μηνών. Μόνο 18 μήνες προβλέπει αυτός ο κώδικας διοντολογίας σε σχέση με το αν μπορεί κανείς να πάει να γίνει λομπίστας μετά τη θητεία του. Έχουμε όμως 36 τουλάχιστον περιπτώσεις ε, πρώην επιτρόπων που πήγανε σε τέτοια ισχυρότατα γραφεία ή και εταιρείες Bank of America, Goldman Sachs, Volkswagen, ε, είναι ελικρούς. Η Επίτροπος για τα ψηφιακά της δεύτερης Επιτροπής Μπαρόσο πήγε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Uber και έχουμε αναφορές που τις προσυμπογράφουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι. Για άλλον επίτροπο που πήγε στην Goldman Sachs. Ρώσο ο ίδιος. Και επίσης Είπαμε τι γίνεται για αυτά τα τοξικά ομόλογα της κρίσης του 8, τα subprime και σήμερα μετά από 16 χρόνια έχουν πληρώσει την ύφη οι Ευρωπαίοι αυτοί που δεν ξέρουν τι γίνεται και δεν φταίνε κιόλα. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κρίση, πώς θα αντιμετωπίσετε τους υπεύθυνους. Λίγα έχουν γίνει σχετικά και τι γίνεται με την Επιτροπή Διοντολογίας που τίποτα δεν έκανε στον ε, σου για την ε, παραβίαση αυτής της υποχρέωσης ε, εντιμότητας. Απάτη. Εδώ βέβαια η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων. Έχει καταραγωθεί αυτή η αξιοπιστία. Θέλετε να λάβετε κάποια μέτρα μέτρα υποχρεωτικά, περιοριστικά, όσον αφορά ακριβώς τη, την υπόθεση αυτών των υπαλλήλων και τις υποχρεώσεις τους. Είπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απαντήστε ό,τι μπορείτε, ό,τι δεν μπορείτε, μπορείτε να το απαντήσετε εγγράφως αργότερα. Ναι, ναι, είναι κλασικέ οι επιτυχίες που ακούστηκαν. Golden Oldies. Κάθε χρόνο παίζουν αυτά τα hits, αυτές οι επιτυχίε των ερωτήσεων. Βέβαια, αυτό είναι η Επιτροπή Αναφορών, να ασχολείστε με όλα και παραπάνω από όλα. Να σα απαντήσω, τέλο πάντων. Σε ευχαριστώ που είπατε ότι βελτιώθηκε η συνεργασία. Θέλουμε να σας καλύψουμε και ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Και εγώ ίδιος θα δω και να φροντίσω να υπάρξουν ποιοτικέ απαντήσεις της Επιτροπής, απαντήσεις προς τους αναφέροντες. Τώρα, τι γίνεται με τους Ευρωπαίους, τι γίνεται με τους Βρετανούς και τον Brexit. Συμφωνώ ακριβώς με τον κύριο Φερχόφστατ, τον διαπραγματευτή σας. Προσωπούμε τα συμφέροντα των 27 στη διαπραγματεύση για τον Brexit, αλλά βέβαια κανείς, κανείς πολίτης, είτε προέρχεται από 27 χώρες είτε από την Βρετανία δεν θα πρέπει να υποφέρει εξαιτία του Brexit. θα πρέπει να προσθέσουν τα σφαίρα των 3 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είναι στη Βρετανία, αλλά και το εκατομμυρίο των ε, Βρετανών που μένουν στις 27 χώρε. Και οι μένοι και οι δε θα πρέπει να προστατευτούν. Άλλωστε, μέχρι τον Brexit παραμένουν Ευρω... πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υποφέρουν μετά τον Brexit. Άρα Όλα αυτά νομίζω ότι διατυπώνονται και θα ε, δημοσιοποιηθούν και στα συμπράσματα του Συμβουλίου του Σαββάτου. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογικές περιφέρειες και την ανακατανομή τους. Γίνεται αυτό σε πολλές χώρε και αυτό άλλωστε γίνεται παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη. Είναι και το θέμα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αυτό με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια. Πολλές φορές, με δύσκολες συνθήκες. Πολλά έχουμε πετύχει, αλλά τη σημερινή ημέρα και πάλι γίνονται τα εξυλαστήρια θύματα. Και έχουμε τις παραδοσιακές αλλά και νέες μειονότητες. Θα πρέπει άρα να πιέσουμε τα κρατημέλη να έχουν συνέπεια στην πολιτική τους. Μα είμαστε τόσο ξεκάθαροι για τις εθνοτικές μειονότητες, δεν θα πρέπει να κουκουλώνουμε το πρόβλημα άλλων μειονοτήτων και να λέμε ότι αυτές οι άλλες μειονότητες είναι απειλή για την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Κάποιοι πολιτικοί αγωνίζονται σκληρά για τους αδελφούς τους, αλήτρωτους ή άλλο κράτος μέλος, ε, αυτοί ε, ας δείξουν επίσης το ίδιο πάθος όσον αφορά το να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Ε, αυτό είναι θέμα το οποίο σηκώνει συζήτηση. Συμφωνούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλές φορές και με τον Όρσα για τις μειονότητες. Και αυτό προσωπικά θα με απασχολήσει. Και με ενδιαφέρει γιατί με τη σημερινή πολιτική συγκυρία στην Ένωση οι μειονότητες πάρα πολύ εύκολα γίνονται στόχος, εξελαστήριο θύμα, ε, είναι ευάλωτες. Και ποια είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μειονότητα. Πάρα πολύ ευάλωτη. Και ενώ τους Ρωμά. Αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Κοινωνικά, πλευράς εκπαίδευσης και η Επιτροπή ασχολείται στα σοβαρά. Τα παιδιά υποφέρουν. Πολύ δύσκολο θέμα. Γιατί αυξάνεται το μίσος για τους Ρωμά. Είναι ο στόχος. Θέλουν κάποιον να καθίσουν το σκαμνί και είναι εύκολο θύμα η Ρώμα όπως κάποτε ήταν οι Εβραίοι. Άρα θα ασχοληθώ ολόψυχα με το θέμα. Αλλά εντάξει και για, για το εκλογικέ περιφέρειες. δικαιώματα των ανηλίκων, κάτι έχω εδώ, σημειώσει. Λέει ένα σωρό χαρτιά εδώ. I'll το χαρτί και θα επανέλθω. Ελπίζω να βοηθήσει εδώ ο συνάδελφος, γιατί δεν το βρίσκω το σχετικό έγγραφο. Τώρα, ο ρόλος της Επιτροπής. Τα έχουμε πει πανελειμμένα με τον κύριο Μαριά. Ελλάδα, θεμελιώδη δικαιώματα. Επιμένει για τα θέματα αυτά ο κύριος ε, Μαριάς. Και πρώτα πρώτα έχω να σας πω ότι τελικά υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Φυσικά υποφέρει πολύ κόσμο στην Ευρώπη. Και είναι ακριβώ το φως στην άκρη του τούνελ. Δεν είναι το φως σαν που έρχεται να σε λιώσει. Ξέρει. Ήδη την απάντησή μου ο κύριος ε, Μαριάς το πριν ρωτήσει, ότι πρόκειται περί συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται περί συμφωνίας με την διεθνή κοινότητα. Δεν θα αμφισβητεί ο κ. Μεριάς ότι έχει καταβάλει ό,τι δυνατή προσπάθεια υπήρχε η Επιτροπή Γιούντερ για να μπορέσει να βγει από το αδιέξοδο η Ελλάδα. Ο κύριος Γιούνκερ, ο κύριος Μοσκοβισή και άλλοι συνάδελφοι πάλι πολλέ φορέ ύψωσαν τον αίσθημά του κατά αυτό που ήθελαν να είναι πιο αυστηροί, πιο σκληροί με την Ελλάδα. Και αυτή την έννοια σα λέω ότι η Επιτροπή είναι φίλη τη Ελλάδο, τη ελληνική κυβέρνηση. Εγώ έτσι το βλέπει και η ελληνική κυβέρνηση από ό,τι ξέρω. Και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι που θα συνεχίσει να σα απασχολεί κύριε Μαριά, αλλά πάλι σα λέω, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα σύμφωνα με τα όσα συμφωνούμε με την ελληνική κυβέρνηση. πολλέ φορέ. υπάρχει δισταγμό του να αυτή η συμφωνία, αλλά εμεί προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο για την Ελλάδα. Τώρα για την ε, μετεγκατάσταση, με ρωτήσατε αν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επί παραβάση. Ε, ακόμα μελετούμε τι θα πρέπει να γίνει τι θα βοηθήσει περισσότερο τους πρόσφυγες που είναι στριμωγμένοι. Ακόμα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα νησιά. Βελτιώθηκε κάπως, αλλά το κρατημέλη κάνουν περισσότερο σε αυτό το μέτωπο από ό,τι πριν. Λίγα κρατημέλη δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι θλιβερό, να το πω διπλωματικά. Αλλά άλλα κρατημέλη όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία κάνουν περισσότερα και όπως θα τους ζητήσαμε. Άρα, να, η ελληνική στην πράξη από αυτά τα κρατημέλη. Και πονάω όταν βλέπω τι γίνεται από λίγα κρατημέλη που κατηγορηματικά αρνούνται να κάνουν οτιδήποτε. Και φτάνουν να λένε στο λαό ότι οι πρόσφυγες είναι κάτι σαν τρομοκράτες. Αυτό με καταραγώνει Δεν ξέρω ότι ε, αυτοί οι πρόσφυγες, οι πραγματικοί πρόσφυγες έτρεξαν να σωθούν από τους τρομοκράτες. Οπότε θα συνεχίσουν να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ότι βοηθάει την κατάσταση. Τέλος πάντων, αυξάνεται την κατάσταση και αυτό είναι καλά μαντάτα. μεταχείριση των παιδιών, την ευημερία των παιδιών, συγκεκριμένα μέτρα. Λέμε, αλλά δεν υπάρχει εδώ αρμοδιότητα της Επιτροπής. Είναι θέμα κρατών μελών. Μας λένε, δεν έχετε αρμοδιότητα, υπάρχει νομικό επιχείρημα το οποίο είναι υπέρ τους. Ευσταθεί. Διαβούλευση συλλογή στοιχείων, όσον αφορά υιοθεσίε. υιοθεσίες. Ε, πολλές χώρες είτε δεν έχουν στατιστικά στοιχεία είτε δεν θέλουν να τα γνωστοποιήσουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας. Έχουν τη σχετική ομάδα εργασίας για τους ανηλίκους. Θα ληφθεί από υπόψη όσον αφορά την ανθεώρηση του σχετικού κανονισμού των Βρυξελών. να υπάρξει όσο γίνεται πιο στεγανές εγγύσεις για τα δικαιώματα των παιδιών. Και υπάρχει ομολογία βέβαια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πολλά επιδέχονται βελτίωση. Μην διστάζετε να μας πείτε το πού χρειάζεται να κάνουμε κάτι. να κάνουμε όπως θέλετε το να εφαρμόσουμε αυτά που έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Θα τα συζητήσουμε με την συνάδελφο, την κυρία Γιούροβα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα η ερμηνεία του άρθρου 51 ή τέλο πάντων η νέα ερμηνεία. Εδώ το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει το το άρθρο 51 ισχύει για τα θεσμικά όργανα και για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 51 ούτως ώστε να ισχύει και σε άλλα πεδία, σε άλλους τομείς πέρα από αυτούς. Δεν μπορεί αυτό να αλλάξει. Τώρα για την συνθήκη του Μαρακές το ΔΕΚ αποφάσισε το Φεβρουάριο ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης η κύρωση της συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αβεβαιότηση. Και νομίζω ότι έτσι προλύνουμε το έδαφος για να κυρώσει το Συμβούλιο την συνθήκη, τη συμφωνία. Το Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει κοινοτικό δίκαιο. Έχουμε δύο νομοθετικέ προτάσεις του Σεπτεμβρίου πέρσι. Και έχουμε τώρα υπό εξέλιξη τον τρίμηρη διάλογο. Ουγγαρία και ο νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση. Αύριο θα το συζητήσουμε αυτό στην Ολομέλεια. Οπότε τώρα δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε θα τα πούμε και στην συνάντηση όλων των επιτρόπων αύριο το πρωί. Προσπάθησα να προετοιμάσω το θέμα. Είχαμε επίσκεψη κάποιου υπουργού, υφυπουργού Ούγγρου να εξηγήσει τη θέση κυβέρνηση. Χθε επίση συνάντησα τον διευθυντή του Κεντρικού Πανεπιστημίου που ήρθε να τα εξηγήσει. Οι νομικοί κοιτάζουν το θέμα από την πλευρά του και θα επανέλθουμε αύριο. Α, για την Ουγγαρία. Επίσης, πάμε στη Ρώμη. Και είπαμε και για το, για την, κοινό μας πεπρωμένο, υπογράψαμε εκείνη τη διακήρυξη. Μετά πάμε στη Βουδαπέστη και πετάμε την, το πυροτέχνημα στόπ στις Βρυξέλλες. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Είναι, δεν υπάρχει καμία συνέπεια μεταξύ της μιας και της άλλης ενέργειας. Είναι πολύ σε επίπεδο θυμικό. Τι είναι αυτό η προσπάθεια χειραγώγηση του πληθυσμού εν ώψη δημοψηφίσματος. Εντάξει, ο καθένα έχει δικαίωμα στην προσωπική του γνώμη, αλλά δεν μπορεί καθένα να κατασκευάζει τα πραγματικά περιστατικά. Είδατε εμεί πώ απευθυνόμαστε στην ε, Ουγγαρία για τα όσα, γίνεται, όσα γίνονται από την κυβέρνηση. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το ότι κάποια πράγματα απλώ είναι αναλυθή. Είναι σαφέ ποιο έκανε τι και έτσι. Θα πρέπει να έχουμε σεβασμό για τον κόσμο και να ενημερώνει το κόσμο σωστά. Νομίζω αυτό είναι το καθήκον μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να αποκαθιστούμε την αλήθεια, να προσπαθούμε. Να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε, ποιος αποφασίζει τι. Άρα να μην έχουμε παρερμηνίες, παρεξηγήσεις. Α, αυτό θα πρέπει να κάνουμε από πλευράς μας. Εκλογές στη Γαλλία, τι να πω. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είδα τις αντιδράσεις πολλών τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους ψήφισαν πολιτικούς που είχαν στάση αντιευρωπαϊκή, που ήταν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οκτώ από τους 11 υποψηφίους του πρώτου γύρου. Οκτώ στους 11 ήταν κατά της Ένωσης. Ε, αυτό πώς να το αγνοήσουμε. Κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει στην κοινωνία. Και να μαζευτούμε εμείς οι φιλοευρωπαίοι και να πούμε «Α, τι ωραία, α, νίκησε ο Μακρόν, βγήκε πρώτος». Καλά, έχουμε και το δεύτερο γύρο των εκλογών, αλλά επίσης το θέμα δεν είναι αυτές οι εκλογές μόνο. Είναι το τι τρέχει στην κοινωνία. Ποιο πριν 900 ετία θα φανταζόταν ότι θα έχουμε τέτοια πράγματα στην ε, Γαλλία κατά τη Ένωση. Αυτό επομένω θα πρέπει να αποτελεί αφορμή προβληματισμού. Ούτε δέχομαι το επιχείρημα ότι για όλα αυτά είμαι εμεί, για όλα αυτά είναι οι αποφάσει των Βρυξελών, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να πείσουμε τον κόσμο για το κοινό μέλλον, το οποίο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με στα ακόμη περισσότερο το έχει κάνει μια ματιά σε όλη την Ένωση. Θα δούμε που είναι οι ακραίοι, που είναι οι οι εθνικιστές δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Το μόνο τους κοινό είναι ότι όλοι μισούν την Ένωση. Την μισούν έντονα και είναι αποφασισμένοι. Ενώ αυτοί που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνουν το ίδιο πάθος, την διαφορετικότητα. Ούτε εδώ, ούτε στα κράτη-μέλη. Να, τι νόημα έχει το να ξανέρθει κανείς κοντά στον κόσμο. Για να δούμε τώρα τι έγινε με τον πρώτο γύρο των εκλογών. Υπήρχαν κάποιες ξεκάθαρες θέσεις. Ο Μακρόν είχε την πιο ξεκαθαρή θέση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνή πολιτική, την μεταρρύθμιση οικονομίας του κράτους κλπ. Και η Μαρίν Λεπέν είχε ξεκάθαρη θέση γι' αυτά. Οπότε αυτό ήταν αιτία να κερδίσουν ψήφους. Να, έτσι θα πρέπει να κάνουμε πολιτική. Και σας το λέω με κάθε ταπεινότητα. Και εγώ από πλευράς του δικού μου κοινωνικού κινήματος που έχει μπροστά σε εκλογικά χαστούκια στις κάτω χώρες και στη Γαλλία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν ο κόσμος θέλει γέφυρες, αυτοί που χτίζουν τις γέφυρες είναι στριμωγμένοι. Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε τώρα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμμετοχή των πολιτών εάν το project πολιτικά είναι ένας τρόπος για να συμβεί αυτό. Πιστεύω πως ναι. στα, για θέματα υπάλληλο δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιοποιούμε πληροφορίες γιατί πρόκειται για διερευνήσεις που κάνουμε για το, ε, το ενδεχόμενο να έχει παραβιαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προσπαθώντας είτε να πείσουμε ε, εκείνων που το έχει παραβιάσει να αλλάξει τακτική ή να ξεκινήσουν μια διαδικασία επί παραβάση. Έχουν ξεκινήσει ορισμένε ε, επίσημε διαδικασίε επί παραβάση για τι οποίε ενημερώνουμε με δελτία τύπου και ε, με άλλου τρόπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέματοφύλακα των συνθήκων και όπως το ποδόσφαιρο, κανείς δεν αγαπάει το διαιτητή. Αλλά δεν μπορεί κανείς να έχει ένα παιδοσφαιρικό αγώνα χωρίς διαιτητή, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αγορά χωρίς κάποιον να φροντίζει για την ε, εύρυθμη και αρμονική έτσι, εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα καταφέρνει, περνάμε στον ανώτερο, αν θέλετε, διαιτητή, το δικαστήριο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπω εγώ τα πράγματα και ίσως έτσι θα έπρεπε να παρουσιάζουμε και τα πράγματα στους πολίτε μας. Η βελτίωση της πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών πιστεύω ότι είναι και αυτή ένας τρόπος ε, μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών. Αναφέρθηκα και στην αρχή. Πράγματι, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιωθούν ε, όσον αφορά τις επιδόσεις τους, τον τρόπο τον οποίο ανταποκρίνονται στις διάφορες αναφορές. Ε, αν το ζητάει και η Επιτροπή Αναφορά του Κοινοβουλίου, ευχαρίστως να το επαναλάβω, γιατί πράγματι είναι στο μέσο στον οποίο χρειάζεται βελτίωση. Τουρκία. Θα διαπιστώσετε ότι όσον αφορά το δημοψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι διεθνείς παρατηρητές του ΟΑΣΕ και αργότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, στην, ε, της επόμενης εβδομάδας, πάνω στην Ολομέλεια, θα γίνει και η συζήτηση για την Τουρκία. Χρηστή διοίκηση. Τι στηρούμε αυτές τις αρχές. Θεωρώ ότι θα έλεγα μάλλον ότι ένα από τα ζητήματα που έρχεται και επανέρχεται είναι η υπόθεση Μπαρόσο, το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι. Θα έχετε διαπιστώσει ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει υποβάλει ορισμένες προτάσεις για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των revolving doors, των υπαλλήλων της Επιτροπής που πηγαίνουν στον τομέα των lobbyist και πίσω συγκεκριμένου κανόνες κανόνε, όπω για παράδειγμα να μην μπορεί κανεί να αναλάβει μια επαγγελματική θέση με αρμοδιότητε σχετικέ με την προηγούμενη ε, θέση που είχε στην Κομισιόν. Η... Ο χρόνο cooling off, ο χρόνο κατά τον οποίο δεν μπορεί κανεί να αναλάβει τέτοιε θέσει, να πάει ε, στα δύο χρόνια για του επιτρόπου και στα τρία χρόνια για τον πρόεδρο τη Επιτροπή. Το συζητούμε αυτό ω ενδεχόμενο, ω πρόταση. Ε, Όμω σε ορισμένε περιπτώσει, πέραν από του δεοντολογικούς κανόνες, εν τέλει, χρειάζονται και πολιτικά πρόσωπα τα οποία να έχουν ευθυκρισία. Αντιλαμβάνονται τι κάνουν. Είδα τις αντιδράσεις των πολιτών στην υπόθεση Goldman Sachs. Ο πρόεδρος Γιούνκερ έθεσε το θέμα στην Επιτροπή Διοντολογίας η επίσημη απάντηση της Επιτροπής Διοντολογίας ήταν ξεκάθαρη, δηλαδή έκανε το έργο της αυτή η Επιτροπή, αλλά ιδιαίτερα δεδομένων, δεδομένης της ιστορίας, του ιστορικού, του, του, του, τοπιών της Goldman Sachs, ε, για να το θέσω πάρα πολύ ευγενικά, σε καμία περίπτωση δεν βοήθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η επιλογή του κ. Μπαρόσου. Γιατί ακόμα και αν κανείς δεν έχει άμεση ευθύνη, δεν εκπροσωπεί πλέον το θεσμικό όργανο, έχει, ε, αντικατοπτρίζονται οι επιλογές του στην εικόνα αυτού του οργάνου. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με, τους, με τον κανονισμό των υπηρεσιακών, τις διαδικασίες που ακολουθούνται πριν από την πρόσληψη ενός ατόμου, για την, την επίσημη εξέταση που γίνεται για το αν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Τώρα, για τους πιο συγκεκριμένους ανθρώπους που αναφέρατε σε, υψηλό, σε υψηλές θέσεις της Επιτροπής δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω ποιους, ε, σε ποιους αναφέρεστε. Δεν γνωρίζω συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πρόσωπο που εργάζεται στην Επιτροπή αξίζει ένα σεβασμό της προσωπικής του ακαιρεότητας, αν, εκτός αν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, Πάντως η διεθνής διαφάνεια, η μη κυβερνητική οργάνωση θα συμφωνήσει μαζί μου, έχει διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς είναι από τις πρώτες θέσεις του τομέα της διαφάνειας. Τώρα, υπάρχει το ζήτημα τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στου κανόνε για τη διαφάνεια. Θα πρέπει να ακούσουμε τη δικιά σα ε, θέση. Είναι ξεκάθαρο πλέον πώ κινούνται τα μέλη τη ε, Επιτροπή και η υψηλόβαθμη αξιωματούχη τη Επιτροπή. Ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει αντίστοιχου κανόνε διοντολογία για τους δικούς του υψηλόβαθμου αξιωματούχου. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, είχα να πω από την δικιά μου την πλευρά. Ελπίζω να απάντησε σε όλε τι ερωτήσει. Η Πρόεδρος να έχουμε χρόνο για ακόμα ένα γύρο ε, συζήτηση. Ναι, ένα λεπτό ερωτήματα. Ο κύριος Κόλλιντς πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλές ε, αναφορές σε σχέση με την εσωτερική αγορά, σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και αυτές έχουν παραμείνει ανεκτές για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να λάβουμε ενημέρωση ε, είτε για την πρόοδο είτε για το εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του παραβάση. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ τους για να αντιμετωπίζουν τις διάφορες ανησυχίες των πολιτών που τους εκφράζονται σε Αυτές οι αναφορές λοιπόν έχουν υποβληθεί σε εμάς και ε, ως προσφυγές στην Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα ξεκίνησαν και οι διαδικασίες επιπαραβάση. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το τι, ε, έχετε, τι βήματα έχετε λάβει από την πλευρά σας για να μας ενημερώσετε, για να ενημερώσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαδικασίες που παραβάση την προηγούμενη χρονιά. Κυρία Σακοράφ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τον κύριο Επίτροπο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη και ουσιαστική θα έλεγα ενημέρωσή του. Ε, οι ερωτήσεις που είχα να κάνω έχουν καλυφθεί ήδη βεβαίως. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας διαβεβαίωσε ότι ο γνώμονάς τους θα είναι η διασφάλιση των των Ευρωπαίων πολιτών και πολύ σύντομα θα δούμε καταγεγραμμένα όλα αυτά. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα τη Ελλάδα και τι ερωτήσει που έβαλε ο κύριο Μαριά, δεν ξέρω τι είδου συζήτηση έχει ξανακάνει με τον κύριο Μαριά, αλλά θέλω να κάνω κάποιε μικρέ μικρές παρατηρήσει πάρα πολύ σύντομε. Όσον αφορά το θέμα του προσφυγικού, που στην Ελλάδα είναι ένα θέμα θα έλεγα, από τα φλέγοντα θέματα, διότι ε, η χώρα μας ε, μέσα σε αυτή την κρίση καλείται να σηκώσει το βάρος που δεν ε, τολμάει να σηκώσει ολόκληρη η Ευρώπη. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Επίτροπο, πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί η Ελλάδα μέσα στην κρίση που περνάει να σηκώσει αυτή την, τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σωστά και σοβαρά πάνω στο θέμα των, της προστασίας και της φιλοξενίας των προσφύγων ή θα πρέπει κάποια στιγμή θέλω να μου το πει αυτό, πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει εκείνα τα μέτρα που θα όφιλε να πάρει ε, απέναντι στα κράτη τα οποία δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ε, όπως κάνει για άλλες περιπτώσεις. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, όσον αφορά το θέμα του χρέους και της ε, επιβολής των μνημονίων στη, στην Ελλάδα. θα διαφωνήσω πάρα πολύ μαζί του, διότι τυχαίνει να είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από την πρώτη μέρα της κρίσης. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον τρόπο που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο, η επιβολή των νόμων και ο τρόπος που έγινε στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν αρμόζει σε κοινοβούλια να, να περνάνε τέτοιου είδους νόμοι, ε, οι μεταρρυθμίσεις που γίνανε, και πάλι θα ρωτήσω, έχει κανόνες ή δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, όταν ε, φροντίζουν να, ε, να διασφαλίσουν την ασυλία των μελών του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή του, του φορέα εκείνου ο οποίος ξεπουλάει κατά δική μου άποψη την ελληνική δημόσια περιουσία. Τελειώνω πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Ή να φροντίσουν την ασυλία των τραπεζιτών οι οποίοι φταίνε για την κρίση κατά ένα μεγάλο μέρος. Την ίδια στιγμή δεν φροντίζουν για τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν, δεν φροντίζουν να εφαρμόσουν το ελάχιστο. Ποιο είναι το ελάχιστο, αυτό που, που, που προσπαθούσαμε και να πούμε από την πρώτη στιγμή. Κύριοι, σε, σε ένα δάνειο έχουν και οι δύο υποχρεώσεις. Και ε, θα πρέπει να δεχτούμε και την ευθύνη αυτών των δύο. Και των δανειστών και των δανειζομένων. Δεν ελέγχθηκε ποτέ και δεν ελέγχθηκε ποτέ το χρέο, κυρία Πρόεδρε, ω οφείλει από τον κανόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσει. Γιατί δεν ελέγχθηκε ποτέ το χρέο τη Ελλάδο. Πώ δημιουργήθηκε. Υπάρχει κανόνα συγκεκριμένο το άρθρο 247 που λέει ότι οι χώρε αυτέ που βρίσκονται σε διαδικασία τέτοια θα πρέπει να ελέγχουν το χρέο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ε, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τιρμερμαντς, δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη σε σχέση με την πρωτοβουλία πολιτών. Το βασικό είναι το εξής. Είναι η συνέχιση, η συνέχεια. Εάν μετά από μια απλή δύσκολη διαδικασία οι, οι προτάσεις των πολιτών δεν οδηγήσουν πουθενά, Δηλαδή, εάν η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο δεν υποχρεούνται να αντιδράσουν, τότε δεν έχει νόημα να ρωτούμε τους πολίτες και να προσπαθούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους. Δεύτερον, απογοητεύομαι όταν σας ακούω να λέτε πως δεν πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 51. Γνωρίζετε πως το άρθρο 51 καταρτίστηκε κυρίως λόγω της πίεσης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας. Πιστεύω πως τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Κατανοώ ότι θέλετε να το εξαλείψετε. Αλλά τουλάχιστον επιτρέψτε μια ανοιχτή ερμηνεία του. Τουν αντίον τα κράτη-μέλη μπορούν να μποϊκοτάρουν τη χάρτη, τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρέντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, έχουμε αναφορές που αφορούν τον Brexit. Και το χειρότερο για τους πολίτες είναι η αβεβαιότητα. Και πολλές φορές δίνεται εντύπωση η Κομισιόν ότι παροξύνει αυτή την ε, αβεβαιότητα. Πρώτα-πρώτα, για ποιο λόγο. Λόγω των διαπραγματεύσεων. Και αναρωτιούνται οι Ευρωπαίοι. Γιατί θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να δοθεί κάποια απάντηση. Είδατε με τον Τιτανικό τι έγινε. Μα τι θα γίνει, δεν, πρέπει να περαμηθούμε των συμφερόντων του κόσμου. Είδατε πώς πήγε 9 μήνες, άλλοι 3 μήνες, τώρα τραβάει το πράγμα. τι θα κάνουμε. Τελικά, τι, τι θα προστατεύσουμε, ποιον θα προστατεύσουμε. Πρόκειται να πάμε εκεί να συζητήσουμε κατά αυτή την περίοδο με τους Βρετανούς ή να τους καλέσουμε εδώ για να τα πούμε. Είναι πολύ λεπτό, δύσκολο θέμα, πολιτικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Σντάνοκα και κατόπιν ο κύριος Βίλαντ Παρακαλώ να είστε πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Πρέπει να φύγει ο Τον Ιούνιο θα συζητήσουμε το τι γίνεται με τα πολιτικά δικαιώματα σε σχέση με το Brexit σε Λατονίκη, σε Εστονία έχουμε πρωτοβουλία πολιτών με 20.000 υπογραφέ σχετικά και η κατάσταση έχει μείνει αμετάβλητη από την ε, προσχώρησή μα. Παρά όλε τι συστάσει, Θα ήθελα η Επιτροπή να ασχοληθεί στα σοβαρά. Να σας δώσω ένα χειρίδο που έχω για το πρόβλημα αυτό για να το αποφετηθείτε. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μου είναι σαν το πρόβλημα που υπάρχει για τους Ευρωπαίους στη Βρετανία και Βρετανούς στην ε, Ευρώπη. Έγιναν ενθαγενείς αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πήγαν από τη μία σοβιτική Δημοκρατία ε, σε άλλη. Δηλαδή σε κάποια βαλτική χώρα που δεν τους αναγνώριζε κάποια δικαιώματα. Δεν αναγνώριζε τόσο πάντων τα ίδια διώματα σε όλους. Ευχαριστώ και ο κύριος Βίλαντ. Κύριε Επίτροπε, τα τελευταία χρόνια η εικόνα των αναφορών άλλαξε. Έχουμε την πρωτοβουλία πολιτών, το διαμεσολαβητή, τις αναφορές, τη συμμετοχή των πολιτών που προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα από κοινού να οξύνουμε και να διαχωρίσουμε περισσότερο τα διάφορα εργαλεία μεταξύ τους και να καταστήσουμε τις διαφορές σαφή στον, στον πολίτη. Στην πρωτοβουλία πολιτών, εν μια πρωτοβουλία είναι επιτυχία, επιτυχής, δηλαδή συγκεντρώσει επαρκή αριθμό υπογραφών, τότε θα πρέπει να υπάρχει και η συνέπεια να πρέπει να αντιδράσουμε. Πιστεύω πως πρέπει να πούμε σαφώς πως μια πρωτοβουλία είναι πρωτοβουλία. Και επίση να μπορούμε να πούμε πω για κάποια πράγματα δεν υπάρχει πολιτική πλειοψηφία. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, χαιρετίζω πολύ αυτό που είπατε για την περαιτέρω ένταξη συμμετοχή του Συμβουλίου καθώς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που δεν είναι υψηλής πολιτικής, αλλά εκνευρίζουν το πολίτη στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και θα ήθελα να διαχωρίσουμε περισσότερο πού μπορεί να υπάρξει κάποια συνέχεια εκ μέρους της ε, Κομισιόν και πού ρητός δεν θα υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας όσον αφορά τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα η κίνηση μιας διαδικασίας επί παραβάση δεν έχω αριθμούς σχετικά με αυτό. Πρέπει να το κοιτάξω να δω σε ποιους τομείς υπάρχει κάτι σχετικό. Με το που θα το μάθω θα σας ενημερώσω. Μόλις αποκτήσω τις πληροφορίες. η Ελλάδα βρίσκεται μόνη της με την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Πιστεύω πως η όλη ιδέα που βρίσκεται πίσω από το κατασκεύασμα του κανονισμού του, Λονδι... του Δουβλίνου συγγνώμη, είναι πως η χώρα της πρώτης άφηξης αναλαμβάνει τον ρόλο Τη υποδοχή και τη καταγραφή των προσφύγων, αλλά όταν καταρτίστηκε ο κανονισμό του Δουβλίνου δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς πως το άχθος αυτό θα επιβαρύνει μόνο ένα ή δύο κράτη-μέλη. Και αν κοιτάξουμε τι γίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και την Ιταλία, ήταν εντελώς άδικο. Πως τόσα πολλά άλλα κράτη-μέλη είπαν έρχονται τόσο πολλοί σε εσά, αλλά έχουμε το Δουβλίνο, πρόβλημά σας. Και αυτό έγινε επί χρόνια και αυτό οδήγησε βρήκε το δρόμο του προς την πολιτική. Κάποια δεν μπορούμε πια άλλο μόνοι μας. Αλλά δεν επήλθε κάποια αντίδραση. Γι' αυτό και κατανοώ τη στάση αυτή. Αν προσπαθεί κανείς επί χρόνια να πάρει μια απόκριση, μια απάντηση, ενώ υπάρχει μια τόσο ανισόρροπη κατάσταση στις αφήξεις. Αλλά από τότε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Ελλάδα, πιστεύω, βίωσε πολύ αλληλεγγύη μέσω ευρωπαϊκών ταμείων, μέσω προστασίας των συνόρων πολλά έγιναν, Πολύ αλληλεγγύη επιδειχθήκε. Ε, εκεί που υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης ακόμα είναι στον τομέα της μετεγκατάστασης. Έχει εγκριθεί, αλλά τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότερο αυτό που υποσχέθηκαν. Και δεν είναι μόνο το ότι λίγα κράτη-μέλη δεν έκαναν τίποτα, αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη υστερούν πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που υποσχέθηκαν όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων που μετεγκαθίστανται. Υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις στο θέμα. Τίποτα δεν έχει επιβληθεί στα κράτη-μέλη. Μπορούν να επιλέξουν τα ίδια. Μπορούν να κάνουν ελέγχους ασφαλείας. Μπορούν να κοιτάξουν το υπόβαθρο των ανθρώπων αυτών. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι που έχουν αποκεφαλίσει άλλους και δεν θα αποκεφαλίσουν άλλου στα κράτη-μέλη. Και λυπούμε πάρα πολύ που κάποιοι πολιτικοί στα κράτη-μέλη το μεταχειρίζονται σαν να είναι μια επιβολή αυτό είναι εντελώ άδικο. Όσον αφορά τη μετεκατάσταση, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Κάποια κράτη-μέλη αποτελούν λαμπρό παράδειγμα, αλλά πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την κατάσταση. Αλλά δεν δέχομαι τη θέση πως η Ελλάδα έχει μείνει μόνη της. Ιδίως στα νησιά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη όντως και κάποιες φορές επίσης τους καταβλισμούς στην υπηρετική χώρα. Αλλά έχουμε επιληφθεί του ζητήματο τώρα και όσον αφορά την οικονομική στήριξη, όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει αλληλεγγύη προ την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση με την Τρόικα και τα μνημόνια, ήδη είπα ότι είχα να πω σχετικά με αυτό. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Μπορείτε να φανταστείτε οποιοδήποτε άλλο κράτο μέλος να χάνει το 1 τέταρτο του εθνικού του πλούτου και δεν είστε ένα από τα πιο πλούσια κράτη-μέλη. Φανταστείτε τι σημαίνει η απώλεια του ενός τετάρτου του εθνικού πλούτου. Βέβαια μπορούμε να αρχίσουμε μια μακρά συζήτηση για νομικά επιχειρήματα, αλλά σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει η απώλεια του ενός τετάρτου του εθνικού πλούτου μιας χώρας. Και τα δεινά που περνάει ο ελληνικός πληθυσμός, ναι, είναι δύσκολα, αλλά πιστεύω πως υπάρχει φως στην άκρη του τόνου του τούνελ. Όσον αφορά την πρωτοβουλία πολιτών, δεν πρέπει να δημιουργούμε υπερβολικές προσδοκίες ναι, η πρωτοβουλία πολιτών πολλές φορές είναι όπως είναι. Είναι μια πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Εάν αναφέρεται σε ζητήματα της αρμοδιότητός μας, τότε πρέπει να πάρουμε θέση. Μας αναγκάζει? Όχι. Αλλά μας αναγκάζει να εκφέρουμε άποψη να προβούμε σε μια αντίδραση στις πρωτοβουλίες των πολιτών. Δυστυχώς, πολλές πρωτοβουλίες που έγιναν μέχρι σήμερα δεν ακολούθησαν τις προδιαγραφές της συνθήκης και του κανονισμού. Τώρα προσπαθούμε να διευρύνουμε την ερμηνεία, το έκανα πρόσφατα, με τμήματα μιας πρωτοβουλίας επειδή στο παρελθόν όταν ένα τμήμα μιας πρωτοβουλίας δεν ενέπιπτε στο προβλεπόμενο πλαίσιο, την απορρίπταμε εξ ολοκλήρου. Τώρα, αν μπορεί να καταχωρηθεί εν μέρη, θα το κάνουμε. Και το δικαστήριο μας διόρθωσε σε μια πρωτοβουλία. Γι' αυτό και τώρα εξετάζουμε τα πράγματα με μεγαλύτερη ακρίβεια και είμαστε πιο ανοιχτοί απέναντι σε εξέλιξεις, αλλά αυτό που είπε ο κύριος Βίλαντ, ναι, ισχύει. Δεν πρέπει να δημιουργούμε υπερβολικές προσδοκίες για τις ε, πρωτοβουλίες πολιτών. Δεν πρόκειται για ένα νομικό εργαλείο. Είναι ένα νομικό εργαλείο, αλλά δεν είναι νομοθετικό εργαλείο. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας το έχει η Κομισιόν και το νομοθετικό δικαίωμα έχουν οι σύνομοθέτε. Ενώ η πρωτοβουλία πολιτών δεν ανήκει σε αυτά. Το 54, το άρθρο 54 είναι μέρο τη συνθήκη μα. Μπορεί να μην σα αρέσει, αλλά δεν συνομιλούμε για τροποποίηση των συνθήκων επί του παρόντο. Και όσο δεν μιλούμε για κάτι τέτοιο, η Κομισιόν πρέπει να σεβαστεί τη συνθήκη. Και αυτό λέει το 54. Η εφαρμογή του χάρτη απόκειται στα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ο ορισμός που εφαρμόζουμε. Όσον αφορά τον χρόνο των διαπραγματεύσεων για το Brexit, αυτό είναι απορρέει από τη διατύπωση του άρθρου 50. Πρέπει να περιμένει κανείς την τυπική ειδοποίηση και στη συνέχεια η όλη διαδικασία κινείται. Ο Μισελ Μπαρνιέ ήταν πολύ ξεκαθαρός για τη σημασία αυτού και ο χρόνος για τη διαπραγματεύσεις είναι πολύ περιορισμένος αν σκεφτεί κανείς την περίπλοκη φύση τους. Και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε στους πολίτες επί του παρόντος και πιστεύω πως πρέπει να το καταστήσουμε σαφές. Επίσης πως τα δικαιώματα των πολιτών βρίσκονται πάνω στην ημερήσια διάταξή μας. Το ζήτημα της ανηθαγένειας στην ε, Εστονία μου είναι γνωστό από τη δεκαετία του 90. Αποδέχομαι ευχαρίστως το έγγραφο που μου παραδώσατε. Μιλήσατε για την μηδενική επιλογή. Η μηδενική επιλογή ήταν δυνατή. και στη Λιθουανία, παραδείγματο χάρη, αλλά η κατάσταση στη Λιθουανία ήταν εντελώ διαφορετική. όσον αφορά τις σχέσεις εντός του έθνους σε σχέση με την Λετωνία και την Εσθονία. Οι χώρες αυτές θεσπίζουν προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ιθαγένειας και οι γνώσεις για τη γλώσσα, για τη χώρα είναι προϋποθέσεις και σε άλλες χώρες. Αλλά και πάλι θα μελετήσω πολύ προσεκτικά το έγγραφο και θα απαντήσω μετά. Οπότε πιστεύω πως απάντησα την ερώτηση επίσης για την πρωτοβουλία πολιτών. Πιστεύω πως αυτά είναι όλα που μπορώ να κάνω για σας σήμερα. Φοβούμαι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαρίστως να ξαναέρθετε. Ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα, συναδελφοί, έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη πριν το μεσημεριανό διάλειμμα. Είναι η 510 σχετικά με τη διασπάθηση χρηματοδότησης. Ο αναφέρον δεν βρίσκεται εδώ, αλλά έχουμε εδώ τον κύριο Όλες Νόβιτς. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, από τη συνάδελφη είναι δύσκολο να κάνει κανείς αυτή την ε, παρέμβαση μετά την ε, ομιλία του Αντιπροέδρου και το γεύμα. Τώρα πρόκειται για ε, χρηματοδότηση η οποία έχει έρθει από το, περιφερειακό, το, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εδώ ο υπεργολάβος είχε την υποχρέωση να εκτελέσει έργα πέραν από την αρχική τιμολόγηση του έργου και ε, αυτό δεν είχε ε, δηλωθεί στον δικαιούχο, χρεοκόπησε. Ε, περίπου 100 άτομα έχασαν την δουλειά τους. Ξετάσαμε το ζήτημα αυτό ήδη από το 2013 στο πλαίσιο προσφυγής και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με το εθνικό δίκαιο. Δηλαδή ότι δεν είχε παραβιαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο όσον αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες, αλλά το αστικό δίκαιο της χώρας ε, όσον αφορά τις ε, συμβάσεις. Το αναφέραμε αυτό στην επιστολή μας pre-closure letter προς τον προσφεύγοντα και η υπόθεση έκλεισε το 2015. Τώρα, πρέπει να δούμε το ζήτημα γενικότερα όσον αφορά τις οδικές τις συμβάσεις για αυτοκινητοδρόμους στην ε, Πολωνία. Το 2008 έως το 2012 η κατάσταση ήταν ε, κάπως ιδιόμορφη. Ο δικαιούχος ζητούσε να γίνουν δεκτές συμβάσεις οι οποίες ήταν υποτιμολογημένες. Και υπήρχε τέτοιο τύπου εξαναγκασμός από τους ε, εργολάβους προς τους υπεργολάβους τους. Τέτοιου τύπου είναι η περίπτωση που συζητούμε. Υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και γενικότερα, για το γενικότερο θέμα, λοιπόν, οι πολωνικές αρχές ανέλαβαν να ε, τηρούν τις υποχρεώσεις τους γενικότερα μιλώντας για τις δημόσιες προμήθειες. Αυτό ήταν η επιδείξη της Επιτροπής, δηλαδή, να κάνουν αυτό το πράγμα οι πολωνικές αρχές. Και πράγματι, το 2012 άλλαξε η νομοθεσία Προστατεύοντα καλύτερα τα δικαιώματα των εργολάβων σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης φροντίσαμε ε, να γίνει πιο ορθή μεταγραφή της οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις στο εθνικό δίκαιο. Έλαβε λοιπόν νομοθετικά, ε, νομοθετικά ε, μέτρα η Πολωνία, βελτιώνοντας τη διαχείριση των των δημοσίων συμβάσεων. στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υποχρεώσαμε τις διαχειριστικές αρχές να εξυγχρονιστούν, να βελτιωθούν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τέτοιου τύπου ε, συμβάσεις. Όσον αφορά για παράδειγμα τις, ε, των προστέρων, ε, τους ελέγχους εκ των προτέρων, εκ προτέρων ζητήσαμε να υποβάλλονται πλέον οι στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να ολοποιήσει το δικό έργο. με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε όλα τα πετούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι αυτή η κατάσταση, αυτή, αυτό το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί. Δεν υπάρχουν πια ε, ε, υποψήφοι ανάδοχοι οι οποίοι να κάνουν προσφορές υπερβολικά χαμηλές. Και ε, όλα αυτά τα βήματα μας οδηγούν στο να είμαστε σίγουροι ότι με τη νέα προγραμματική περίοδο όλα είναι εντάξει. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη αναφορά, η συγκεκριμένη αναφορά αφορά το εθνικό δίκαιο, γιατί η Πολωνία είναι εκείνη που είναι ε, αρμόδια να λύσει το πρόβλημα αυτό, μιας και το ε, ταμείο αυτό βρίσκεται υπό ε, επιμερισμένη διαχείριση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει και να λύσει μια διαμάχη η οποία έχει ανακύψει μεταξύ της διαχειριστικής, της πολωνικής διαχειριστικής αρχής και του εργολάβου, του αναδόχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας περιέγραψα ήδη, ασχολήθηκε με τα δομικά προβλήματα, με τα συστημικά προβλήματα της χώρας έκλεισε το, ο φάκελος το 2015 παρόλα αυτά παρακολουθούμε, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Ο κύριος Γιώργη. Θέλω να μιλήσω πρώτος γιατί έχω μια σύνδεση που αρχίζει τώρα. Κάποιοι πέφτουν από εκείνη την κατάσταση στην Πολωνία, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε νομικό, σε δικαστικό επίπεδο στη χώρα. Αλλά τέλο πάντων αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε και αυτό σας προτείνω είναι ότι να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να στείλουμε μια επιστολή στις πολωνικές αρχές. Να του ζητήσουμε να μα εξηγήσουν τι κάνανε να διορθώσουν την κατάσταση. Ίσως αυτό να γίνει ε, και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πριν κλείσει η αναφορά. Γεια. Είμαι τη ίδια άποψη με τον συνάδελφο, αλλά θα ήθελα να το δώσω στην Ειδική Επιτροπή. Είναι η ελευθερία των συμβάσεων στα κράτη-μέλη, αλλά είναι και ευρωπαϊκά χρήματα που ξοδεύουμε εδώ και δεν μπορεί τώρα λόγω της συμβατικής διαμόρφωσης να έχουμε τμήματα που αποφελούν τρίτους. Τώρα έχουμε να κάνουμε με υπεργολάβους. Αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, αλλά πρέπει να διασπεραλιστεί πως όταν ο υπεργολάβος κάνει τη δουλειά του, ο κύριος ανάδοχος να μην τσεπώνει τα χρήματα, να κηρύσει πτώχευση και στη συνέχεια αυτός που έκανε τη δουλειά να μην πάρει τα χρήματα. Και δεν είναι δυνατόν στο τέλος να μένει, να ξεμένει αυτός που έκανε τη δουλειά. Αυτό με εκνευρίζει, με εξοργίζει. Και όλο αυτό λόγω των, της νομικής διαμόρφωσης της σύμβασης. Η Κομισιόν ασχολήθηκε με το ζήτημα, αλλά μπορούμε να ξαναρωτήσουμε από το Κοινοβούλιο. Όταν ξοδεύουμε ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή όταν επενδύουμε σε υποδομές, επίσης τονώνουμε την οικονομία. Δηλαδή συμφωνώ με τον συνάδελφο. Η ίδια Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Στο μέλλον τα πράγματα ίσως να είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον αναφέροντα. Η Πρόεδρος. Καλώς. Πέτρο, δεν νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έχουμε υπερβεί τα χρονικά όρια μας. Τέλος πάντων, αυτό που προκύψει από τον Γιάννη Γαλαδιοψή είναι ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή αναφορά. Επίσης, ότι θα πρέπει να απευθύνουμε μια επιστολή στις πολωνικές αρχές για να ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Αυτά θα γίνουν. Και να δούμε. Γιατί όντως τα εθνικά δικαστήρια ή τέλος πάντων κάποιοι εθνικοί φορείς έχουν αρμοδιότητα σε τέτοια ζητήματα. Αυτό και θα κάνουμε, θα στείλουμε αυτή την ε, επιστολή και θα κρατήσουμε και την αναφορά. Ευχαριστούμε τους ε, μεταφραστές, που τιμόνων, τους διερμηνείς γιατί δούψαν ένα τρίλεπτο παραπάνω.